Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι περιμένετε για το σημείο 24. Η κυρία Μακοβέη δεν είναι διαθέσιμη, αλλά αντικαθίσταται από την κυρία Στίβενς. Αλλά τώρα έχουμε ζητήσει την ομιλία για τους διερμηνείς μέχρι να φτάσει. Θα διακόψουμε για πέντε λεπτά. για να μπορέσει να αντικαταστήσει καταλληλώς και η κυρία Στίβεν στην κυρία Μακοβέη να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών και θα συνεχίσουμε με το σημείο 24 για τη Σέγγεν. Αν περιμένετε λοιπόν για το σημείο αυτό, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή 5 λεπτών και θα ξαναρχίσουμε για να μπορέσει η κυρία Στίβενς να αντικαταστήσει την κυρία Μακοβέη. Μόλις έρθει η ομιλία θα ξεκινήσουμε. Το πολύ 5 λεπτά. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση συνάδελφοι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πρόκειται για την εφαρμογή των ε, εναπομεινόντων περιορισμών ε, του κεκτημένου Σέγγεν σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Η κυρία Μακοβέη είναι η συγγήτρια, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στίβενς που την αντικαθιστά. Στις 18 Ιανουαρίου το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει για την σκοπούμενη απόφαση να αντιθέσει εφαρμογή ενεπομείνοντες ε, διατάξεις του συγκεκριμένου Σέγγεν σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ο στόχος της απόφασης του Συμβουλίου είναι να έρθουν οι περιορισμοί που παραμένουν για τη χρήση του ΣΥΣ από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και η δυνατότητα να ε, καταχωρήσουν θεωρούνται ε, ειδοποίησης ε, του ΣΥΣ ε, για τους σκοπούς της άρνησης της εισόδου ή της παραμονής και της εκτέλεξης τέτοιων ειδοποιήσεων που εκδίδεται από τα κράτη-μέλη. Κύριε Μακοβέη είναι η συγγήτρια της έκθεσης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας το Συμβούλιο έστειλε στο Κοινοβούλιο αναφερμένη εκδοχή αυτού του σχεδίου απόφασης. Οι κύριες αλλαγές είναι μια παραπομπή στο άρθρο 25 της Σύμβασης Έγκεν που αφορούν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μεταξύ τους και σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη Σέγγεν και δεύτερον μια ημερομηνία θέση εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου, του σχεδίου απόφασης. Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν να ακούσουμε την παρουσίαση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου από την Προεδρία, να έχουμε ένα feedback από την Κομισιόν και κατόπιν να έχουμε παρουσίαση της ε, έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης από την κυρία Στίβενς που αντικαθιστά την κυρία Μακοβέη. συμφωνείτε λοιπόν, θα προχωρήσουμε με τις παρουσιάσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σέκοφ, αντί για την κυρία Μενκόβα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Στίβενς, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, επιτρέψτε μου, εκ μέρους του Συμβουλίου, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης, για την απόφαση του Συμβουλίου, για να τεθούν σε ισχύ ένα από μήνες διατάξεις του κεκτημένου Σέγγεν που σχετίζονται με το ΣΥΣ, Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Για το Συμβούλιο, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να ενδυναμωθεί περαιτέρω η συνεργασία του ΣΥΣ μεταξύ των κρατών μελών. Παρουσιάσατε το σχέδιο της απόφασης, το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι η απόφαση ακολουθεί τη συμφωνία ε, για το σύστημα εισόδου-εξόδου και προβλέπει ότι το σύστημα εισόδου-εξόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να τεθεί σε λειτουργία από κράτη-μέλη που δεν πληρούν στο 100% το κεκτημένο Σέγγεν. Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις στο σύστημα εισόδου-εξόδου για τα κράτη που δεν εφαρμόζουν πλήρω το κεκτημένο Σέγγεν. Η πρώτη προπόθεση, ο πρώτο όρο είναι η πλήρη ε, αξιολογήσει Σέγγεν, να έχουν υλοποιηθεί δηλαδή επιτυχώ οι αξιολογήσει. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία το έκαναν αυτό πριν κάποιο καιρό. Η δεύτερη προπόθεση είναι να εφαρμόζονται οι διατάξει του κεκτημένου Σέγγεν ε, σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών για τι θεωρήσει. Η απόφαση αυτή ήδη ισχύει και εδώ έχουμε την τρίτη απόφαση να διασφαλίσουμε ότι οι διατάξεις του ΣΥΣ τίθενται σε εφαρμογή για τις δύο χώρες. Το Συμβούλιο έχει ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα για να προετοιμάσει το σχέδιο της απόφασης, προκειμένου να υλοποιηθεί ο τελευταίος όρος που θα επιτρέψει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να εφαρμόσει το να εφαρμόσουν το ΣΥΣ χωρίς ε, εναπομείνοντες περιορισμούς, έτσι όπως λέμε στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της απόφασης του Συμβουλίου 2010, κάθετος 265 Ευρωπαϊκή Ένωση, του 2010 όπως σας είπα, για την εφαρμογή των διατάξεων ε, σε, του κεκτημένου Σέγγεν στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η απόφαση θα επιτρέψει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να αξιολογήσουν ε, τις καταχωρήσεις για την είσοδο άλλων κρατών μελών και να λάβουν τις ε, απαιτούμενες δράσεις, δηλαδή να αρνηθούν την είσοδο ε, σε άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπουν στο χώρο Σέγγεν. Ταυτόχρονα, αυτά τα δύο κράτη-μέλη θα μπορούν να κάνουν καταχωρήσεις στο σύστημα και θα μπορούν αυτές οι απαγορεύσεις εισόδου να εκτελούνται από άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην Κομισιόν. Ο κύριος Μαρκέ έχει το λόγο. Η κυρία. Ευχαριστώ. Βιλκλάχο λέγομαι. Καλημέρα στην κυρία Στίβενς και στα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν γενικά καλωσορίζει την απόφαση, καθώς ε, θα συμπεριληφθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία στη συνεργασία Σέγγεν. Επίσης, είναι ένα σημαντικό μέτρο για την βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την απόφαση αυτή, μετά την υιοθέτησή της, η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα μπορούν να ε, κάνουν ε, καταχωρήσεις άρνησης εισόδου στο ΣΥΣ και τα άλλα κράτη-μέλη θα βλέπουν αυτές τις καταχωρήσεις ε, της άρνησης εισόδου από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα μπορούν ε, να αναλάβουν δράσεις στα εξωτερικά σύνορα δυνάμει των καταχωρήσεων αυτών. Θέλω να αναφέρω ότι από τεχνική σκοπιά έχουν γίνει προετοιμασίες ε, από το Ιουλίσα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για να αρχίσει να λειτουργεί αυτό η λειτουργία. Έχουν ε, ολοκληρωθεί δοκιμές από το Ιουλίσα και η Βουλγαρία και η Ρουμανία σε ε, ένα περιβάλλον τεστ μπόρεσαν να δημιουργήσουν αυτές τις καταχωρήσεις στο σύστημα. Έτσι λοιπόν όλα είναι έτοιμα προκειμένου η απόφαση αυτή να τεθεί σε εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά. Να αναφέρω ότι από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν προτιμότερο αν ε, το μέτρο αυτό αποτελούσε συνέπεια της ε, άρσης ε, των ελεγχών στα εσωτερικά σύνορα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν οι έλεγχοι αυτοί και έχουμε ακόμη αρκετές διατάξεις του κεκτημένου Σέγγεν που δεν εφαρμόζονται πλήρως για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς περαιτέρω ολοκλήρωση, όμως όπως ανέφερα θα ήταν προτιμότερο αν Κάτι τέτοιο αποτελούσε συνέπεια της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του κεκτημένου Σέγγεν και, του, ε, και της πλήρους άρσης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Μάλιστα, ευχαριστώ τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με την κυρία Στίβενς που θα μιλήσει εκ μέρους της κυρίας Μακοβέη. Παρακαλώ. Uh, thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω εκ μέρους ε, της κυρίας Μακοβέη, που δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί γιατί είναι άρρωστη. Χαίρομαι που εγώ την αντικαθιστώ για το συγκεκριμένο θέμα. Ε, η απόφαση άρρη απομείνοντες περιορισμού για τη χρήση του ΣΥΣ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αυτοί οι περιορισμοί αναφέρονται στην υποχρέωση άρνησης εισόδου ή διαμονής ε, σε υπηκός τρίτος χωρός, ε, αν υπάρχει καταχώρηση που έχει ε, εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος για τους ε, σκοπούς ε, της άρνησης ε, της της διαμονής εκδίδονται τέτοιε καταχωρήσεις. Όταν υιοθετηθεί η απόφαση του Συμβουλίου, οι έλεγχοι που γίνονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα εξωτερικά σύνορα και στην επικρατεία τους θα είναι πιο αποτελεσματικοί. Τα δύο κράτη-μέλη θα μπορέσουν να εκδώσουν καταχωρήσεις ΣΥΣ προκειμένου να αρνηθούν την είσοδο ή την παραμονή και ταυτόχρονα να εκτελούν αυτές τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει από όλα κράτη-μέλη. Η την παραμονη και ταυτοχρονα να εκτελουν αυτες τις καταχωρησεις που εχουν γινει απο άλλα κρατη μελη η συνεισφορα στην ασφάλεια της Ένωσης θα αυξηθεί, ιδίω αν τέτοιε καταχωρήσεις βασίζονται σε απειλή στην δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια ή στην εθνική ασφάλεια. Η εισηγήτρια καλωσορίζει την απόφαση του Συμβουλίου και μας υπενθυμίζει ότι και η Βουλγαρία και η Ρουμανία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ε, σε επιχειρήσεις παρακολούθησης στον Ευξηνοπόντων αλλά και στο Δούναβι που είναι στρατηγική διάδρομη, είναι ανοιχτή σε παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία και αποτελούν ε, τροτά σημεία. Ταυτόχρονα και οι δύο χώρες ε, ήταν σημαντικές συνεισφορέ σε επιμελητιακή υποστήριξη ε, στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Συνοριακής και Εκτοφυλακής. Αυτό αποτελεί σημαντική εξέλιξη προκειμένου η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Επιπρόσθετα, αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενδυναμωθεί η καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατίας η συγγήτρια συνιστά το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του Συμβουλίου χωρίς ε, τροπολογίες για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν ταχύτατα στην υιοθέτηση της απόφασης. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι Δευτέρα Μαΐου και εδώ στη ΛΥΜΠΕ η ψηφοφορία θα γίνει στις 24 Μαΐου. Προβλέπεται στις 24 Μαΐου. Ευχαριστώ, Χέλγα. Τώρα, ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Κουέλιο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το 2011 είχα την τιμή να είμαι ο εισηγητής του σώματος για την ε, ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν. Αλλά ακόμη και σήμερα δυστυχώς η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό το χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας. Και επανειλημμένα έκτοτε έχω τονίσει. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έκαναν σωστά αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν, αλλά η ομοφωνία στο Συμβούλιο δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν. Αυτό είναι άδικο. Και καταδεικνύει τα προβλήματα που προκαλεί η ομοφωνία. Χθες, την πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του χωρού Σέγγεν, της οποίας είμαι εισηγητής, είπαμε ανεπιφύλακτα. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία πρέπει απευθείας και χωρίς επιφυλάξεις να, είναι, να καταστούν πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν. Σήμερα αυτό το σχέδιο έκθεση είναι άλλο ένα βήμα ακριβώ για να ενταχθούν αυτέ οι δύο χώρε σε ένα ουσιώδε τμήμα του Σέγγεν. Το SIS. Ελπίζω ότι εύκολα και ταχύτατα θα συνενέσουμε για να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί για τους ελέγχους στα σύνορα. Όπως λέει η συγκήτρια, αυτά τα δύο κράτη-μέλη θα συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερο στην ασφάλεια του χώρου Σέγγεν. Αλλά δεν υποφελούνται από την άλλη όψη του νομίσματος περισσότερο ελεύθερη κυκλοφορία. Το ΕΛΚΑ θα συνεργαστεί με την εισηγήτρια και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει πλήρης ένταξη στο χώρο Σέγγεν, όχι μόνο στο SIS της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Αυτός πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν σαφέστατο νομίζω. Ο κύριος Κουαϊού και η κυρία Φιέλνερ η κυρία Φαγιόν είναι η συγγήτρια, έχει το λόγο. Λοιπόν, θα διαβάσω το κείμενο που προετοίμασε ο σκιώδης μας, ο κύριος ε, Στάνισοφ. Ευχαριστεί τον εισηγητή που εργάζεται για αυτό το θέμα. Τον Οκτώβριο το Συμβούλιο ενέκρινε μία απόφαση για να χορηγηθεί στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία παθητική πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωσης για τις ε, βίζες. Μαζί με το θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αυτές είναι οι δύο τελευταίες διατάξεις του κεκτημένου του Σέγγεν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν αρθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι στα σύνορα. Είναι προϋποθέσεις για να ε, ενταχθούν και στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που θα αρχίσει να λειτουργεί το 20. Τώρα λοιπόν αυτές οι δύο χώρες θα έχουν και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις πλήρους συμμετοχής ε, στο Σέγγεν. Όμως στο Συμβούλιο δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση, άρα δεν μπορούν να υποφεληθούν από την άρση των συνόρων στα... των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Έχουν περάσει περίπου 7 χρόνια από τη στιγμή που ε, το Συμβούλιο είχε πει ότι και νομικά και τεχνικά σε όλους τους τομείς ε, του κεκτημένου Σέγγεν οι δύο χώρες ήταν έτοιμες. Όμως μόνο τώρα βλέπουμε ένα μικρό βήμα, όχι λόγω του ότι πληρούν τα κριτήρια, τα κριτήρια αλλά επειδή αυξάνονται συνεχώς οι πιέσεις για περισσότερη ασφάλεια, πολύ συχνά εις βάρος ε, των πολιτικών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ασφάλεια χωρίς να σέβεται τις εγγύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ασφάλειας χρειάζεται κοινή δράση. Πρέπει να υπάρχει σωστή στάθμιση μεταξύ ασφάλειας και ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το νομικό πλαίσιο είναι παρκώς ρωμαλαίο και όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το να υπάρχουν αόρατα σύνορα μεταξύ κρατών μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα από τα πιο απτά και σημαντικότερα επιτεύγματα της Ένωσης εξυπηρετεί μόνο την υπονόμευση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Να μπορέσουν αυτές οι δύο χώρες να ε, εποφελούνται από το SIS χωρίς ε, περιορισμούς είναι ένα καθυστερημένο βήμα, παρόλα αυτά καλοδεχούμενο και στηρίζω πλήρως την εισηγήτρια στην εργασία της. Αυτά λέει ο Σεργέη Στάνιουσερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι και οι δύο ε, πολύ σωστά περιγράψατε τη θέση της Επιτροπής μας. Ο κύριος Αντάμοφ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το θέμα του Σέγγεν είναι πολύ ρεπτό για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Γι' αυτό να μην ξεχνάμε ότι τον Ιούνιο του 2011, στις 9 συγκεκριμένα Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο κατέληξε ότι ίσχυαν όλες οι προποθέσεις για τα χερσαία και εναέρια σύνορα, τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών, την προστασία των δεδομένων, τα θαλάσσια σύνορα, τις προξενικές ορίσεις, ότι όλα αυτά, όλα αυτά τα κριτήρια πληρούνται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Παρ' όλα αυτά, Ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει καταλήξει το Συμβούλιο σε μια τελική απόφαση, γιατί δυστυχώς πρέπει να ληφθεί ισότιμα από όλα τα κράτη Σέγγεν. Αυτό είναι ιδιαίτερα άδικο. Γιατί η Βουλγαρία και η Ρουμανία προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ευχαριστώ τον κύριο Κάρλος Κουέλιου για τη στάση του και για τον κόπο του για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ που θεωρείτε ότι και οι δύο αυτές χώρες πρέπει να ενταχθούν αμέσως στο χώρο Σέγγεν. Θα υποστηρίξουμε το σχέδιο απόφασης γιατί θα συμβάλλει στην άρση των ε, τελευταίων περιορισμών για την χρήση του SAS από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της ομοκρατίας και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Άνταμο. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Οπότε. Κύριε Στίβενς, θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Θέλετε να κάνετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Όχι. Όχι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να αναφέρω Κάναμε μια συνάντηση με το ίδιο e Λίσα, αλλά χωρίς επαρκή συμμετοχή δυστυχώς για τις προπαρασκευαστικές ε, εργασίες τεχνικής φύσης. του ΕΣΑΕΣ. Αλλά δυστυχώς ε, δεν είχε ευρεία συμμετοχή γιατί συνεδρίαζε παράλληλα η ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία αλλά ετέθησαν και εκεί σε αυτή τη συνάντηση αυτά τα θέματα. Πώς θα βοηθήσουμε να υπάρξει αυτή η πρόοδος. Θέλει κανείς να πει τίποτα άλλο γι' αυτό. Ωραία. Ωραία. Αυτά προς αυτό. Κυρία Στίβες, δεν θα προσθέσετε τίποτα. Ναι, με συγχωρείτε. Για το ίδιο e Λίσσα. Από ό,τι κατάλαβα από τις, ε, τους συνεργάτες της κυρίας Μακοβέη, όλοι έχουν ήδη ολοκληρωθεί, έχουν προετοιμαστεί. Και χθε έγιναν και κάποιε δοκιμές και πήγαν καλά. Πολύ καλά. Απλώς για ενημέρωση. Νομίζω ότι πρέπει να το ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Κλείνουμε το θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα στο 24. Ερώτηση για γραπτή απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 8ης 11 για τον Ιταλικό νόμο που λέει ότι τα στοιχεία των τηλεπικοινωνιών πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για 6 χρόνια. Να, αποθηκεύονται. Είναι ερώτηση της κυρίας Σοφ Είναι άλλη μια ερώτηση που δεν απαντήθηκε εν Την υπέβαλε η κυρία Ιντφελντ. Η προθεσμία για να ληφθεί απάντηση ήταν η 15η πρώτου τρέχοντος αλλά δεν υπήρξε απάντηση. Και γι' αυτό η συντάκτρια ζήτησε σας παρακαλώ φεύγουν να μην κάνουν φασαρία. Λοιπόν, η συγκήτρια ε, ζήτησε το θέμα αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξή μα με βάση τον, το άρθρο 130 παράγραφος 5. Εν τω μεταξύ η Επιτροπή απάντησε στην ερώτηση. Αλλά παρόλα αυτά η συντάκτρια θα ήθελε να ασχοληθεί η Επιτροπή μα. και να ακούσει και την προφορική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σοφή, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Διστάζω λίγο πρέπει να ομολογήσω. Γιατί εδώ συζητάμε για ένα σοβαρό πολιτικό θέμα και ο μόνος ευρωβουλευτής στην αίθουσα Εντάξει, υπάρχουν αξιωματούχοι της Επιτροπής, λένε ωραία 10 λεπτά, θα υποστώ την οργή της κυρίας Ινφετφέλτ και τελείωσε. Αλλά κανένα άλλο. Έτσι θα αντιμετωπίζουμε σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Τι κίνητρο υπάρχει έτσι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίρνει στα σοβαρά τις γραπτές ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν εμεί οι ίδιοι δεν είμαστε εδώ παρόντε. Οπότε ειλικρινά εγώ δεν θεωρώ ότι έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Το τελικό κοινοβούλιο με τον πιο έτσι κρυφό τρόπο ποτέ Εκτός από την περίπτωση του iCloud στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς πέρασε. Πέρασε λοιπόν το Ιταλικό Κοινοβούλιο μια νομοθεσία για την αποθήκευση δεδομένων για έξι χρόνια. Μα είναι υπερβολικό. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό, πήραμε βέβαια πολύ αργά την απάντηση, τι λέει, λέει, δεν μας αφορά, είναι θέμα των εθνικών αρχών, εμείς ετοιμάζουμε έτσι καλώς νομοθεσία για να νομιμοποιήσουμε αυτή την πρακτική. Αυτή είναι η απάντηση. Και εδώ είμαι μόνο εγώ, άντε και εσείς, βουλευτές και κανένας άλλος στην αίθουσα. Μα δεν είναι αυτός τρόπος, πρόεδρος. Κοιτάξτε για το θέμα της λογοδοσίας και το μηχανισμό λογοδοσίας, το θέμα της παρουσίας μάλλον. Υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα εδώ, γιατί υπάρχουν πολλές συνεδριάσεις που γίνονται συγχρόνως επικαλύψεις. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα δηλαδή όσον αφορά την παρουσία των Ευρωβουλευτών στις συνεδριάσεις. Πάντως, αν μη τι άλλο, θέλω να στηρίξω το μηχανισμό, παρόλο που μερικές φορές καταλήγει σε τέτοια κατάσταση ελάχιστης παρουσίας Ευρωβουλευτών, γιατί μη τι άλλο υπάρχει η διευκόλυνση να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το άρθρο 130 δεν ξέρω αν δεν νομίζω ότι λες ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το μηχανισμό. Είναι σημαντικό να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ βάσει αυτού του άρθρου και να μας απαντάει. Η κυρία Χετφέλτ. Μα δεν είναι ευρωβουλευτές εδώ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε ένα μέσον που αναργαλείο που ονομάζεται γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Και τι κάνει με αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίποτα στις ε, αδιάφορες ερωτήσεις που δεν έχουν μεγάλη σημασία, απαντάει αμέσω. Στις άλλες δεν απαντάνε στις πιο σοβαρές. Μέχρι να επιμείνεις και να ξαναεπιμείνεις και μέχρι να μην έχει πια νόημα. Έτσι θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους αυτούς μας. Δεν λέω ότι θεωρώ ότι χάνω το χρόνο μου μιλώντας σε ένα αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα βαθύ πολιτικό ζήτημα. Έχουμε δώσει τόσες μάχες για την αποθήκευση δεδομένων. Πριν από καιρό χρόνια κράτησε μια δικαστική ε, περίπτωση γι' αυτό. οι Ιταλικές αρχές τι λένε, δεν τους ενδιαφέρει, τέλος πάντων. Πρόεδρος. Ναι, Έχετε εκνευριστεί, το καταλαβαίνω. Το ερώτημα είναι, λέει κυρία Ινχιτφέλτ, πώ θα το αντιμετωπίζουμε. Δεν πρόκειται για τι διαδικασίε, δεν πρόκειται τι ώρα μέσα στην ημέρα βάζουμε το ένα θέμα ή το άλλο. Είναι πόσο σοβαρά ε, παίρνουμε ένα εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να λογοδοτούν σε εμά η το αλλο ειναι ποσο σοβαρα παιρνουμε ενα εργαλειο που εχουμε στη διαθεση μα προκειμενου να λογοδοτουν σε εμα η ευρωπαικη επιτροπη και οι χώρε μέλη. Στις δικαστικές αποφάσεις, αν η Επιτροπή οι χώρες μέλη συστηματικά ε, αδιαφορούν για τις αποφάσεις του δικαστηρίου, εμείς πώς αντιδράμε. Λέμε δεν μας νοιάζει. Αυτό είναι το σημερινό διακύβευμα. Λοιπόν, επιμένω να επανέλθει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και όχι μόνο σε σχέση με αυτήν την ε, κοινοβουλευτική ερώτηση, αλλά γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοιες ε, καταστάσεις. Πρόεδρος, το σκεφτόμουν όσο μιλούσατε, πράγματι μπορεί υπό διαφορετική μορφή να ξαναμπεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ναι. Αυτή η ερώτηση, έτσι, να ξαναμπεί στην ημερήσια διάταξη σύντομα, αυτό λέτε. Και οι συντονιστές όμως να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον αυτό το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας των γραπτών ερωτήσεων. Ωραία. Εσείς και εγώ θα συνεχίσουμε το διάλογο, όμως μια που είμαστε οι δυο μας μόνο εδώ. Ωραία, το σημειώνουμε. Αυτό θα ξαναμπεί στην ημερήσια διάταξη. Ναι, λέει η κυρία Χετφέλτ. Θέλω στην πρώτη συνάντηση της Λίβε μετά από αυτήν να μπει πάλι στην ημερήσια διάταξη. Έτσι κι αλλιώ το πολιτικό σα ζήτημα το θέσατε και μεταφέρθηκε και στο διαδίκτυο, εφόσον η συνεδρίασή μα μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ωραία, σα ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναμπεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης και στι συνεδρίες των συντονιστών. Συναδελφοί, σημείο 25 τώρα. Προβλέπονταν για τις 10 και 30. Μου λένε να διακόψουμε 15 λεπτά και να επανέλθουμε στις 10 και 30 για να συζητήσουμε για την Eurojust. Τι θέλει να απαντήσει η Επιτροπή. Αντιλαμβάνεστε ότι έκλεισε το θέμα, δεν μπορούμε να επανέλθουμε. Το τελειώσαμε, το κλείσαμε. Πραγματικά θέλετε να επιστρέψουμε. Θα ήθελα να αντιδράσω, επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, για τα σχόλια όσον αφορά την υποχρέωση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λογοδοτεί και να απαντάει σε αυτές τις προφορικές ερωτήσεις. Επί της ουσίας θα απαντήσω την επόμενη φορά, εντάξει. Ειλικρινά θέλετε να επανέλθουμε. Είσαστε σίγουρος. Σας δίνω τη δυνατότητα να μην έχοντας κλείσει αυτό το θέμα. Είσαστε σίγουρος ότι θέλετε να επανέλθετε. Γι' αυτό το βάλαμε επειδή δεν απαντάτε έγκαιρα. Τώρα έρχεστε εδώ, το κλείνουμε το θέμα, δεν σας είδα. Και τώρα πραγματικά είσαστε σίγουρος, θέλετε να επιχειρηματολογήσετε γι' αυτό. Εγώ θα σας συμβούλευα να μην το κάνετε, η κυρία Χετβέλτ. Μέχρι τώρα όλα ήταν πολύ φιλικά, αλλά αν μας μεταχειρίζονται έτσι δεν θα είμαστε πια τόσο φιλικοί. Ας πάμε για καφέ καλύτερα. Μιλάνε συγχρόνως ο Πρόεδρος και εκπρόσωπος της Επιτροπής. Συμβουλεύω να κλείσουμε το θέμα εδώ, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνώ, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ωραία, επαναρχόμαστε στις 10.30. και we'll get started. Um, I'll, I'll, I'll explain everything and I'll actually say that we could do it again. Okay, colleagues, um, so we're going to... Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με το σημείο 25, τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Συνεργασία στην Ποινική Δικαιοσύνη, τη Eurojust. Θα ήθελα να καλωσορίσω σήμερα τον κύριο Χάμρεν, τον πρόεδρο του Eurojust, να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση. Είναι καινούριο στο καθηκοντά ο κύριος ε, Χάμραν σχετικά. Ε, είχαμε κάποιες ε, συναντήσεις σε σχέση με την ουσία των καθηκόντων της Eurojust. Ήταν εξαιρετικές οι συνεδριάσεις αυτές, οι συναντήσεις αυτές και πραγματικά πιστεύω ότι θα παράσχει μια ευρωστηγησία στην Eurojust. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σε σχέση με τη συμμετοχή σήμερα. Ήταν κάπως ασυνήθιστη ημέρα. Νομίζω ότι ε, κάπως εξαντλούνται δυνατότητα στις επιτροπές. Ε, είχαμε ε, εδώ συμμετοχή <laughs> σε συγκεκριμένα τμήματα της συνεδρίασης. Είναι και web stream τη συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ε, βέβαια, Ελπίζω ότι θα ήταν ε, περισσότεροι βουλευτές ε, παρόντες. Ε, θα ήθελα να τα πω αυτά για να μην νιώθετε απεσιόδοξα. Ευχαριστώ την κυρία Σίπελ που είναι εδώ. <laughs> Είναι ίσως ένα από τα μέλη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ίσχυρα και σε προηγούμενες συνεδριάσεις είχαμε μέλη που συμμετείχαν πολλά. Βέβαια, μας παρακολουθούν και από το διαδίκτυο θα κάνετε μία παρουσίαση σε εμά, όπως σας είπα. Καταγράφετε, αλλά ξέρω ότι θα ξανάρθετε σίγουρα, σύντομα, όταν θα είναι και πιο πολλοί βουλευτές παρόντες. Είχαμε συνεδριθεί και στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθεί και ο Eurojust να επικοινωνεί. Θα σας ακούσουμε και στην παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το ένθερμο καλωσόρισμα. Είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα και χαίρομαι που θα σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση το 2017, για το 2017, όταν η συνθήκη του Μάστρεκτ ε, εισήγα για την δικαστική ε, και αστυνομική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει πριν 25 χρόνια, τότε ήταν πολύ διαφορετική η καιρή. Τότε το έγκλημα ήταν πολύ πιο περιορισμένο στα εθνικά σύνορα από τη σήμερα και οι ε, εισαγγελείς ε, ε, συνήθως χρησιμοποιούσαν απρόβλεπτες διπλωματικούς διάβλους, έστελναν επιστολές ετοιμάτων μέσω των κεντρικών αρχών. Δεν υπήρχε διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών, ούτε θεσμική πλατφόρμα για να αναλύσουμε, να συντονίσουμε τις υποθέσεις με συναδέλφους από όλα κράτη-μέλη. Τα τελευταία 25 χρόνια είδαμε μια τεράστια εξέλιξη στον τομέα της ασφαλείας και της δικαιοσύνης. Η ετήσια έκθεση του Eurojust για το 2017 ε, το απεικονίζει αυτό. Αποτελεί μια συγκεκριμένη απόδειξη για το πόσο μακριά έχουμε πάει τα τελευταία 25 χρόνια. Θα δείτε στην έκθεση συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα και ουσιαστικά έχουν κάνει την Ευρώπη πιο ασφαλή. 25 χρόνια εξακολουθούμε να έχουμε 28 κράτη-μέλη με διαφορετικές ε, δικαιοδοσίες, με διαφορετικούς κανόνες που σχετίζονται με τις ποινικέ διαδικασίες. Επίσης, έχουν και διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με το παραδεκτό των ε, αποδείξεων. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι εισαγγελείς χρειάζονται την Eurojust να είναι πιο αποτελεσματικοί, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Eurojust για το συντονισμό των ερευνών, για την ε, σύραξη, όταν υπάρχει σύγκρουση δικαιοδοσιών και για τη συλλογή αποδείξεων με έναν τρόπο που να είναι παραδεκτός στα εθνικά δικαστήρια. Πέρσι ε, το έργο της ε, Eurojust ε, κατέγραψε πάνω από 4.000 υποθέσεις, σχεδόν 4.500 εισαγγελείς, δικαστές και αστυνομικοί από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και όχι μόνο, ήρθαν στο Eurojust για να πετύχουν αποτελέσματα. Ένας από αυτούς ήταν ένας εισαγγελέας από την Άπολη, από την Ιταλία. Θα ε, ήθελα να σας εξηγήσω πώς αναπτύχθηκε η υπόθεσή του και τι σήμαινε η εμπλοκή της Γιούρουτζας για τη δική του υπόθεση. Επομένως, ε, πάμε στην Άπολη, 2015, η Ιταλική Αστυνομία ε, κατάσχει ένα φορτίο ναρκωτικών, ανακαλύπτει την εισαγγελία ότι οι υποπτήσεις συνδέονται με την Ιταλική Γκομόρα, την Ιταλική Μαφία. Οι εισαγγελείς στην Νάπολη έρχονται σε επαφή με τη Γιούρουτζας, θα αναζητούν βοήθεια να στη βοήθεια ο αγγελέα ε, και μα ε, ρωτούν από πού παίρνουν τα ναρκωτικά οι υποπτοί, συνεργάζονται ε, με άλλε εγκληματικέ ομάδε σε άλλε χώρε, υπάρχουν άλλοι εισαγγελεί που να ερευνούν του ίδιου υπόπτου ή τι ίδιε εγκληματικέ ομάδε που να δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω τη Eurojust αποκαλύπτεται σύντομα σύνδεσμοι με μια ισπανική εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται σε ελαφρεμπόριο ναρκωτικών και εκβιασμού και ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Ε, ε, χρησιμοποιούν την περιοξενοσύνη τη Eurojust για να συσταθεί μια κοινή ερευνητική ομάδα από εδώ και πέρα. Έτσι θα εργάζονται οι αρχέ Πέρσι η Eurojust υποστήριξε 200 κοινέ ερευνητικέ ομάδε. Ε, μαζική αύξηση από, το από δύο ομάδε το 2002. Αυτό μα δείχνει την τεράστια εξέλιξη που κάναμε στον τομέα τη δικαιοσύνη και τη ασφάλεια. από το 1993. Επίση, σε σύντο χρόνο, συνεόμαστε με την ποινική ε, δραστηριστή Γερμανία Αγγελής. Από τρει χώρε ε, τώρα εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Έχουν συμφωνήσει σε μια κοινή στρατηγική για το πώ θα αποφευχθεί η σύγκρουση δικαιοδοσιών και συζητούν ε, διάφορα νομικά προβλήματα που σχετίζονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψη ή με ευρωπαϊκά ερευνητικά εντάλματα, ευρωπαϊκά εντάλματα έρευνας. Κατόπιν αυτών φτάσαμε σε ένα κρίσιμο σημείο σημείο τον ε, Ιούλιο του 2015 στις 5 Ιουλίου στις 4.30 ε, το πρωί οι εισαγγελείς από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία ε, συναντιούνται στη Χάγη στο κέντρο συντονισμού και μπορούν να έχουν μία ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ε, σε διάφορους ε, τόπους. Ε, έχουμε stand-by των αστυνομικών ή εισαγγελείς, εργάζονται δίπλα-δίπλα οι γυροστές και οι αστυνομικές ομάδες αρχίζουν να εκτελούν τις συλλήψεις, τις κατασχέσεις. Ταυτόχρονα έχουμε σύνομη επικαιροποίηση συνεχώς και όσο προχωράει η μέρα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες. Και νέα στοιχεία λοιπόν, νέες συνδέσεις που εμείς απευθείας καταλήγουν σε δράση. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση συνελήφθησαν 33 άτομα σε τρεις χώρες την ίδια μέρα, 5 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από ένα τόνο ναρκωτικά κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση αυτή είχε τον κωδικό Σάντα Λουτσία και την διάλεξα γιατί ε, βοήθησε ε, η Eurojust με όλες τις δυνατότητες της ε, κέντρο συντονισμού, νομική ανάλυση, κοινή δράση. Αυτά είναι τα σημαντικά και μοναδικά στοιχεία που μπορεί να αξιοποιήσει η Eurojust για μεγάλης κλίμακας και περίπλοκες υποθέσεις. Αλλά και ένα άλλο στοιχείο για αυτή την υπόθεση. Στην αρχή ήταν μια τοπική αστυνομική επιχείρηση, μικρών διαστάσεων νομίζαμε, αλλά τελικά είχε πολλές ε, διεθνείς διασυνδέσεις και μας πήρε χρόνια. Χάρη στο συντονισμό μας που είναι μόνο δυνατό μας στους Eurojust, επιτύχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Όλοι ξέρουμε ότι το έγκλημα δεν σταματάει στα σύνορα ούτε καν τη ε, Ένωση. Γι' αυτό η συνεργασία και με τρίτα κράτη είναι ουσιώδε στοιχείο τη δουλειά μα. Η Eurojust από την αρχή οικοδομεί ένα δίκτυο δικαστικών σημείων επαφή που τώρα περιλαμβάνει 42 τρίτε χώρε και θα επεκταθεί περισσότερο τους επόμενους μήνες. Και στα κτίρια μας έχουμε και ε, τους εισαγγελείς ε, επαφής με τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων το Μαυρογούνιο και οι Ηνωμένες Μία από τις πιο περίπλοκες υποθέσεις που αντιμετώπισε το 2017 ε, ε, ε, ε, αφορούσε έρευνα για θέματα ποδοσφαίρου, για παράδειγμα στήσιμο παιχνιδιών, ε, απάτες, παραγαράξεις εγγράφων και είχε πολλές ε, διακλαδώσεις. Ξεκίνησε από την Ελβετία και είχε διακλαδώσεις στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Και η υπόθεση αυτή τελικά κατέληξε σε μια μέρα δράσης που ήταν ε, συντονισμένη από εθνικούς εισαγγελείς από το κέντρο συντονισμού της Eurojust και ε, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ε, υλικών εγκλήματος αλλά και κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη της ενοχής. Στην Ουγγαρία για παράδειγμα. Σε ένα σημείο στον ε, αυτοκινόδρομο πυροβολείται ένα άτομο, ένας Ούγγρος και φαίνεται ότι είναι Γερμανός ο δράστης. Οι Ουγγρικές αρχές μέσω του κέντρου που είναι 24 ώρες 24 ώρο συνεχώς σε λειτουργία ζήτησαν βοήθεια και θέλησαν να ξεκινήσει να υπάρξει μια εντολή ευρωπαϊκής έρευνας για να γίνει μια έρευνα κατοίκων στην Γερμανία. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι ο ύποπτο είχε δανείσει το αυτοκίνητό του σε έναν συγγενή του στην Αυστρία. Ξεκίνησε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό ένταλμα ε, σύλληψη και ένα νέο ένταλμα ευρωπαϊκής Έρευνα. Αλλάξαμε λοιπόν τη δικαιοδοσία από τη Γερμανία. Μέσα σε δύο ώρες περάσαμε στην Αυστρία. Με ένα νέο ένταλμα σύλληψη και νέο, ε, νέα εντολή έρευνας κατοίκων. Λιγότερο από 24 ώρε μετά το αδίκημα συνελήφθη ο υποπτό. και όλα τα στοιχεία για την απόδειξη συμπεριλαμβανομένου του όπλου ήταν στην κατοχή μα. Αν δούμε την ευρύτερη εικόνα αποτελεσμάτων, θεωρούμε ότι είναι ακόμη πιο εύγλωτα. Ασχοληθήκαμε με 10 υψηλή ορατότητα υποθέσει σε 10 διαφορετικού τομεί εγκληματική δραστηριότητα και βλέπετε τα αποτελέσματα. Χάρη στην Eurojust, οι εθνικέ αρχέ συνέλαβαν 345 μέλη εγκληματικών οργανώσεων και έκαναν πάνω από 300 έρευνες κατοίκων και κατέσχεσαν ε, υλικά εγκλήματος αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καταπληκτικό γιατί σκεφτείτε ότι ο τίσος προπολογισμό μας είναι 37,5 εκατομμύρια. Ακόμη πιο σημαντικό. Η Eurojust βοήθησε τους ανακριτές, τους εισαγγελείς να έχουν επαρκή στοιχεία που να μπορούν να βοηθήσουν σε δικαστικές διερευνήσεις. Το όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας το Κοινοβούλιο συνεχίζει να παίζει ουσιώδη ρόλο. Ως νομοθέτες έχετε συμβάλει στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων δικαστικής συνεργασίας που είναι ουσιώδη στην καταπολέμηση του διαμεθοριακού εγκλήματος. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ε, ε, εντολές παγώματος στοιχείων ενεργητικού ή εντολές ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι έχουμε τους αναγκαίους πόρους για την αρχή του προπολογισμού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ειλικρινά για τη στήριξή σας. Και σας ευχαριστώ γενικότερα. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αυτό είναι το μέλλον της Eurojust για το μέλλον. Είναι η ετήσια αύξηση υποθέσεων που μας απασχολούν. Είναι γύρω στο 10% το χρόνο. Δηλαδή εκατοντάδες νέες υποθέσεις κάθε χρόνο. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό και περισσότερο χρόνο για κάθε υπόθεση. Και τι άλλο βλέπουμε. Ότι ορισμένες φορές δεν έχουμε επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις υποθέσεις. Κάναμε μία σε βάθος μεταρρύθμιση για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και μία αναδιοργάνωση της χρήσης των πόρων μας για να δίνουμε περισσότερη στήριξη στα εθνικά μας γραφεία και στις εθνικές αρχές. Αλλά δεν επαρκούν όλα αυτά, γιατί υποβάλλονται όλο και περισσότερα αιτήματα από τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, το 2019 ζητήσαμε λίγο περισσότερο, πάνω από 41 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρειαζόμαστε αυτά για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, για να μπορούμε να δώσουμε απτή βοήθεια στα κράτη-μέλη, για να χρηματοδοτούμε ομάδες κοινών ερευνών ή για να συντονίζουμε μεγάλες κλίμακας επιχειρήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν να μα στηρίξετε στις επερχόμενες συζητήσει για τον προπολισμό του 19 αλλά και περαιτέρω του 2020 ούτω ώστε η Eurojust να παίξει το ρόλο της να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή τη που είναι η δικαιοσύνη πέρα από τα σύνορα. Σήμερα δεν σας παρουσιάζω μόνο τη Eurojust τη δουλειά μας δηλαδή, αλλά να σας παρουσιάσω και τους 330 αφοσιωμένους συνεργάτες μας. Τα επιτεύγματά μας είναι αποτελέσματα της δικής τους αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς. Όλοι μαζί είμαστε η Eurojust. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα πιο ασφαλές, ένα πιο δίκαιο χώρο. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Λίμπε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τη συνεχιζόμενη στήριξή σας. Ευχαριστώ για την θαυμάσια παρουσία σας. και για τον πολύ άμεσο τρόπο παρουσίασής της. Να απευθυνθώ στο μέλος. Εξαίρετο μέλος. Την Birgit, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση αυτή. Θέλω να επικεντρωθώ σε δύο διαφορετικούς τομείς. Αρχίσατε λέγοντας ότι μετά από, από 25 χρόνια και παρά τη συνεργασία που έχουμε, οι νομικοί κανόνες διαφέρουν μεταξύ των χωρών και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στα αποδεικτικά στοιχεία άλλου κράτους. Το ξέρουμε ότι είναι διαφορετική κατάσταση Στι 28 χώρες. Αλλά ποια είναι ακριβώς αυτή. Πότε μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς. Αυτό είναι που διαφέρει. Είναι το σε τι πράγμα μπορεί να έχουν πρόσβαση αρχές άλλης χώρας. Υπάρχει μια φήμη και δεν φτάνει η φήμη για να ζητήσουν πρόσβαση σε στοιχεία οι αρχές, πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, τι. Μιλήσατε και για την ομάδα και την κοινή ερευνών. Η χρηματική ενίσχυση πάει και εκεί ή υπάρχει άλλη χρηματοδότηση που μπορείτε να δίνετε στις χώρες μέλη για να κάνουν αυτέ τη δουλειά του. Έπειτα λέτε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες περιπτώσεις που χειρίζεστε και ότι ίσω δεν είστε πλήρως εξαπλισμένος για να τα καταφέρετε. Οπότε αυτή η αύξηση και στην ομολογία σημαίνει επίσης ότι υπάρχει και περισσότερη εγκληματική δραστηριότητα διασυνοριακά ή ότι υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση στις χώρες μέλη και σας ζητούν βοήθεια όλο και πιο συχνά. Μπορεί να είναι και τα δύο βέβαια. Η κατάσταση λοιπόν είπαμε στις χώρες μέλη διαφέρει πολύ όσον αφορά τους κανόνες. Μπορεί να χρειαζόμαστε ενίσχυση της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών. Κάποιες χώρες θα έπρεπε να κάνουν περισσότερες προσπάθειες αυτό. Αναφερθήκατε επίσης και στον φόρτο εργασίας της Eurojust. Λοιπόν, οπότε μήπως χρειάζεται περισσότερα χρήματα Eurojust. Η ερώτηση βέβαια δεν είναι τόσο για σας, είναι περισσότερο προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι έτοιμη η Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν περισσότερα όπου χρειάζεται, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρήματα εννοώ, έτσι, περισσότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Και τέλος, ίσως εσείς βέβαια μπορεί να μην επιτρέπετε καν να τοποθετηθείτε από αυτού, η ερώτηση είναι πάλι προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τα χρήματα για τη Eurojust και για όλα τα άλλα που χρειάζονται οι χώρες μέλη και τα ζητούν από την Ευρώπη, η Επιτροπή και το Συμβούλιο σκέφτονται πηγές για τη χρηματοδότηση αυτή. Για τελείως ωραία είναι να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά δεν έχουμε αρκετά περισσότερα χρήματα, παγιδευόμαστε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια σχόλια και ερωτήσεις που είχα. Σε κάποια μπορείτε να απαντήσετε, σε άλλα φαντάζομαι είναι περισσότερο για να απαντηθούν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Λοιπόν, και εγώ έχω ερωτήσεις. Να ρωτήσω κι εγώ, έτσι καλώς δεν θα υπάρξουν άλλες και μετά να απαντήσετε. Συζητήσαμε για διάφορα θέματα και για αυτά που συζητιούνται στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη. Όταν προσπαθείτε να κάνετε μεταρρυθμίσεις στη Eurojust, και τα έχουν ακούσει και νωρίτερα οι συνάδελφοι, παλιότερα, Τι ακριβώς συγκεκριμένα προσπαθείτε να μεταρρυθμίσετε. Τι θα αλλάξει δηλαδή. Γιατί ένα από τα αξιοσημείωτα θέματα είναι ο προπολογισμό, που είναι ελάχιστος δεδομένων των τόσων πολλών δραστηριοτήτων της Eurojust στις διάφορες χώρες. Οπότε είναι ενδιαφέρον Ο προπολογισμό αυτός πρέπει να χρηματοδοτήσει και τις κοινέ ερευνητικές ομάδες σε ένα τόσο δύσκολο πεδίο δράσης. Ποια είναι η προτεραιότητα τώρα. Εσείς δώσατε παραδείγματα με χώρες. Εγώ θα μιλήσω για την Σλοβακία. Πήγαμε στη Σλοβακία πρόσφατα και εκεί ήταν σαφές τι θέλαμε η δικιά μας κοινοβουλευτική, δηλαδή αντιπροσωπεία από την Europol. Αυτό, να υπάρχει κοινή έρευνα, κοινέ ερευνητικές ομάδες που να μπορούν να βοηθήσουν τις σλοβακικές αρχές στην περίπτωση της δολοφονίας του κ. Κιούτσιακ. Θέματα όμως συστημικά για να πάρω αυτό το παράδειγμα πάντα τη Σλοβακία, Θα μπορούσε να αφορά και τη Ρουμανία ή οποιαδήποτε άλλη, το ξέπλυμα χρήματο κλπ. Πώ αποφασίζετε όταν έχετε τόσα πολλά ζητήματα που θα δώσετε την προτεραιότητα. Είδα την ετήσια έκθεσή σας και είδα ότι ασχολείστε με πολλά και διαφορετικά θέματα σε διάφορε χώρε. Πώ τα επιλέγετε όμω, Οπότε πάλι για να επανέλθω στην περίπτωση τη Σλοβακία. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διάφορα τρέχοντα ζητήματα, ε, υπόνοιες που θα μπορούσατε να είχατε παρέμβει από αυτόν. Ε, θέματα δικαστικού σώματος. Έχετε ασχοληθεί με αυτά σε άλλες χώρες, καθυστερήσεις συστημικές που δυσκολεύουν τη δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι αυτά τα θέματα αφορούν αποκλειστικά τη Σλοβακία. Οπότε Ποιε είναι οι προτεραιότητες σας, πώς καθορίζετε μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, θέλετε να ασχοληθείτε με θέματα που προκύπτουν επίκαιρα, εγκληματικές ε, δραστηριότητες. Και τότε δεν ε, έρχονται σε αντίθεση δικές σας οι δραστηριότητες με εκείνες τη Europol γιατί υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα δικαστών, εισαγγελέων. Και μετά υπάρχει η σύνδεσή σας με τους εισαγγελείς. Ξέρω ότι τα χρήματα είναι λίγα. Και για το μέλλον το θέμα του προϋπολογισμού θα είναι πολύ σημαντικό για την Eurojust. Ακριβώς επειδή εξετάζετε τόσα πολλά θέματα και παρεμβαίνετε σε τόσες πολλές υποθέσεις. Η κυρία Σίπελ. Να προσθέσω κάτι. Αναφερθήκατε και στην κατάρτιση. Έχετε κι εσείς μια ειδική μονάδα όπως στη Σίπολ ή πώς γίνεται η κατάρτιση έχετε εσεί τη δική μονάδα ή γίνεται απαλού. Πρόεδρος, να διευκρινίσουμε λίγο αυτό το θέμα που σας είπα της ε, ασυμβατότητας. Πού είναι η διαχωριστική γραμμή, είτε πρόκειται για δικαστές είτε άλλους που δουλεύουν στον τομέα της ασφάλειας και έχετε κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Πώς το αποφασίζετε, το συζητάτε με τους άλλους, το συζητάτε στην Επιτροπή, πώς παίρνετε τις αποφάσεις σας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο φαντάζομαι, αλλά πώς ε, καταλήγετε στην στρατηγική σας δράση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες ως πακέτο. Καταρχήν, να αποσαφηνίσω ότι η Eurojust δεν έχει εντολή ως προς την κατάρτιση την εκπαίδευση. Είμαστε ένας οργανισμός που λειτουργούμε βάσει της ζήτησης. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη που εξακολουθούν να ερευνούν όλα αυτά τα εγκλήματα, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, Και υπάρχει ένα διεθνές, ε, μια διεθνή συνιστόσα στην υπόθεσή τους και αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, νομικά προβλήματα, προβλήματα επικοινωνίας, οικονομικά προβλήματα. Τότε εκούσια παραπέμπουν τις υποθέσεις τους στη Eurojust. Δεν υπάρχει λοιπόν υποχρέωση των κρατών μελών ε, να παραπέμψουν τις υποθέσεις τους στη Eurojust. Αυτές οι υποθέσεις που είναι στην ετήσια έκθεση συνολικά περίπου 2.700 είναι εκούσιες συνεισφορές από τα κράτη-μέλη. Και τους δίνουμε τη βοήθεια που χρειάζονται. Ίσως να είναι ένα νομικό ζήτημα που να προκύπτει από διαφορετική εφαρμογή κάποιου νομοθετικού μέσου ευρωπαϊκού. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει κάποια νομοθετικά μέσα με διαφορετικό τρόπο. Και στην πράξη φαίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε αυτά τα ζητήματα και πρέπει να συζητήσουμε για να βρούμε κάποια λύση και μια ρεαλιστική προσέγγιση για να προχωρήσουμε. Επίσης, μπορεί να έρχουν ε, κάποιες χερσές επιχειρήσεις και θέλουν να συστήσουν κοινέ επιχειρησικέ ε, ερευνητικές ομάδες. Μπορεί να μην έχουν εμπειρογνωμοσύνη ως ε, προς την διαπραγμάτευση μιας τέτοιας ομάδας. Δεν ξέρουν τι να συμπεριλάβουν στη συμφωνία της ερευνητικής ομάδας, δεν ξέρουν ποιε είναι οι απαιτήσει θέλουν παραδείγματο χάρη να συναντηθούν, να παρουσιάσουν την υπόθεση στη Eurojust, να εξηγήσουν την υπόθεση στους συναδέλφους, να προτείνουν μια συμφωνία κοινή ερευνητική ομάδα και να συζητήσουν του όρου, τι προποθέσει βάσει τι οποίε θα βασίζεται η συμφωνία. Έτσι, λοιπόν, αντιμετωπίζουμε πραγματικά νομικά, πρακτικά ζητήματα. Έτσι βοηθάμε τους ε, υπαλλήλου ε, στον κλάδο. Πολλές φορές ε, υπάρχει βούληση από διάφορες χώρες ε, να συνάψουν μια συμφωνία κοινή έρευνα. Αν όμως έχεις μια κοινή ερευνητική ομάδα, τότε οι άνθρωποι θα πρέπει να συνεργαστούν, να συναντηθούν, να ταξιδέψουν και δεν είναι πολύ συχνά έτοιμοι να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες γιατί χρειάζεται διερμηνία, μετάφραση, κάποιος να κλείσει τις πτήσεις. Επίσης χρειάζονται ειδικέ συσκευές ε, που θα σου διασφαλίσουν μια ασφαλή σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ των μέλων της ομάδας. Εδώ λοιπόν έρχεται και παρεμβαίνει η Eurojust, είναι μια ανάγκη αυτή και αυτός είναι και ο λόγος που πραγματικά αγωνιζόμαστε για περισσότερη χρηματοδότηση για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, ο προϋπολογισμός δεν είναι μεγάλος, 37,5 εκατομμύρια. Αλλά από τον προϋπολογισμό αυτό, 1,3 εκατομμύρια επιστρέφεται στα κράτη-μέλη στις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Και βλέπουμε μια αυξανόμενη ζήτηση όπως είπα το 2002 είχαμε δύο ερευνητικές ομάδες, αλλά μετά από 15 χρόνια βλέπουμε ότι η Eurojust υποστήριξε 200 τέτοιες ερευνητικές ομάδες και οι κοινέ ερευνητικές ομάδες ποτέ δεν ασχολούνται με μικρές ή μεσές υποθέσεις. Μιλάμε για πολύ μεγάλες σημαντικές υποθέσεις, τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων. κάποιες υποθέσεις που αφορούν νομοποίηση παράνομων ε, εσόδων, εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία ναρκωτικών ή όπλων, φορολογικές υποθέσεις. Είναι λοιπόν διασυνοριακές εκφύσεως οι υποθέσεις αυτές. Αυτά κάνουμε. Τώρα, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Συνειδητοποίησαμε ότι το προσωπικό μα που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να παράσχει την υποστήριξη, την ιδιοποιότητα στην υποστήριξη που θέλουμε να δώσουμε και εξετάσαμε από κριτική σκοπιά πώς δαπανούμε τους πόρους μας. Έτσι βρήκαμε κάποιους τρόπους πώς να κάνουμε μια νέα κατανομή και πραγματικά να εστιάσουμε σε πραγματική επιχειρησιακή υποστήριξη. Συζητήσαμε την κατάσταση στο σώμα και το σώμα της Eurojust που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια στρατηγική απόφαση ότι πρέπει να κάνουμε νέα κατανομή των πόρων και από τα διοικητικά καθήκοντα να έχουμε περισσότερους πόρους που να ενεργοποιούνται για επιχειρησιακά καθήκοντα. Έτσι βλέπουμε το μέλλον. Θέλουμε να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στην ε, επιχειρησιακή δουλειά, δηλαδή στην υποστήριξη, στη δουλειά επί των υποθέσεων και να επικεντρωθούμε σε νομικά ζητήματα και να παράσχουμε πρακτική υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Σε σχέση με την ερώτηση που αφορά τα 27 διαφορετικά νομικά καθεστώτα, Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε 28 κράτη-μέλη, έχουμε 28 διαφορετικούς νομικούς πολιτισμούς, 28 διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Και μάλιστα σας είπα ήδη ότι οι διάφορε χώρες μπορεί να εφαρμόζουν διαφορετικά τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα, όχι ομοιόμορφα. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε τα πάντα. Δηλαδή, ακόμη και με το μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης, παρόλα αυτά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ε, διάφορες δικονομικές απαιτήσεις. Ε, ας δούμε, τους χάρη, τις έρευνες κατοίκων. Οι έρευνες κατοίκων στην Ιταλία απαιτούν δικαστική έγκριση, το ίδιο και στη Σλοβακία. Όμως, οι απαιτήσει ε, για να δοθεί αυτή η έγκριση μπορεί να διαφέρουν αναχώρα. Εκεί λοιπόν τίθεται το θέμα του παραδεκτού των αποδείξεων, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ό,τι συλλέγεται στην Ιταλία είναι παραδεκτό και σε διαδικασίες δικαστικές στη Σλοβακία. Σε σχέση τώρα με την κατάσταση του προσωπικού στα κράτη-μέλη δεν έχω συγκεκριμένα αριθμιστικά στοιχεία, δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω. για την κατάσταση στη Σλοβακία και σε άλλες χώρες. Όπως είπα, δεν επικεντρωνόμαστε στην κατάρτιση. Πώς βασικά διαλέγουμε το πεδίο των δρασιών μας. Προσπαθούμε να εξαλείψουμε, να φιλτράρουμε, αν θέλετε, τις ίσονος σημασίας υποθέσεις. Νομίζω ότι βάση δικαστικής παραγγελίας. Πώς βοηθάτε τα δικαστικά συστήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κενά και ανησυχίε. Αν υπάρχει δηλαδή τέτοιο αίτημα, τέτοια δικαστική παραγγελία. Νομίζω ότι γίνεται κατόπιν αιτήματος. Επομένως δεν μπορείτε στην πραγματικότητα να παρέμβετε. Ναι, ναι, ακριβώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση οι Σλοβακικές αρχέ σε πρώιμο στάδιο παρέπεμψαν την υπόθεση στην Europol και στη Eurojust. Στις 18 Απριλίου είχαμε μια συντονιστική συνεδρίαση με τους Ιταλούς συναδέλφους στη Eurojust και ήταν παρούσα και η Europol. Έτσι βλέπουμε και το μέλλον μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να συνεργαστούμε και διάφορες χώρες, διάφοροι οργανισμοί να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γιατί μόνο αν συνεργαστούμε όλοι μαζί μπορούμε να επιλύσουμε διάφορα δύσκολα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις διαφορετικές δικαιοδοσίες. Μάλιστα, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση, πολύ καλή ετήσια έκθεση. Ε, πραγματικά βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ε, ε, ουσιαστικά ουσία Eurojust, ουσιαστικά ασχολείται με τις διάφορες ερευνητικές εντολές, με τα εντάλματα έρευνας. Αυτή είναι η καθημερινή δουλειά που έχετε. Και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε και εμείς από τη σκοπιά της λογοδοσίας. Ξέρω ότι θέλετε να διατηρήσετε αυτή την πολύ στενή σχέση με την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τη χαμηλή συμμετοχή. Όμως ε, θα υπάρξει και νέα συνάντηση και θα διατηρήσουμε τις σχέσεις μας στενές. Ε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη. Ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα σε λίγα λεπτά. Dear colleagues, if everyone is... Αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αλλά παρακαλώ, καθίστε. Μια ώρα έχουμε. Αλλά καλό παρακαλώ καθίστε. αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε μια ώρα στη διάθεσή μα μόνο, <coughs> άρα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σημείο 27 τη μέρης της διάταξη, κατάσταση στην Ουγγαρία. Με βάση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17 η Μαΐου 2017. Εξετάζουμε τώρα το σχέδιο έκθεσης. Η συγκίτρια μας είναι η κυρία Σαρτζεντίνη. Έχουμε τον κύριο Πίτερ Ζουχάρτο που είναι ο Ούγγρος Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου. Στις 17 Μαΐου το Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Στην παράγραφο 10 το Κοινοβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή μας να ξεκινήσει τη διαδικασία και να συντάξει έκθεση με στόχο να γίνει ψήφιση, ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να λυθεί δράση κατά της ε, Ουγγαρία με βάση το άρθρο 7 της συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Σαρτζεντίνη ορίστηκε εισηγήτρια στι 11 Ιουλίου 2017. Έκτοτε έχει συνεργαστεί με τους Κιώδης, οι περισσότεροι είναι σήμερα παρόντες, για να προπαρασκευάσει αυτή την έκθεση. Η κυρία Σαρτζεντίνη παρουσίασε τα πορίσματά της ε, για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης στη συνεδρίασή μας στις 12 Απριλίου. Σήμερα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση. να καλωσορίσω και τον κύριο Πίτερ Σουχάρτο που είναι Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας. Λοιπόν, να δώσω απευθεία το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Τζούντιθ Σαρτζεντίνη. Πριν πάρει το λόγο, θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε μόνο μία ώρα για το θέμα. Για να έχουμε λοιπόν διερμηνία μέχρι το τέλος της συνεδρίασης παρακαλώ να τηρήσετε όλο το χρόνο σας. Σας παρακαλώ να μην τον υπερβαίνετε. Κυρία Σαρτζεντίνη, παρακαλώ το πολύ 10 λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε στην έκθεση. Να κάνω και εγώ μια επισκόπηση. Η έκθεση βασίζεται στο άρθρο 83 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου, που λέει ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να κάνει μια ετολογημένη πρόταση καλώντα το Συμβούλιο να δράσει με βάση το άρθρο 7, παράγραφο 1 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον ε, περασμένο Μάιο η Ολομέλεια έδωσε εντολή στη ΛΥΜΠΕ να συντάξει μια έκθεση θεωρώντας, όπως τόνισε, ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία αποτελεί ε, ε, σοβαρή απειλή παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 και γι' αυτό αιτιολογείται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7.1. Χρησιμοποίησα την περίοδο ε, του περασμένου, της περασμένης άνοιξης για να ε, διερευνήσουμε την κατάσταση. Είχαμε καλέσει και την Ουγγρική κυβέρνηση, και είχαμε και μία πλήρη συνεδρίαση των σκιωδών για να ακούσουμε τις εξηγήσει του πρέσβη της Ουγγαρίας εδώ. Ακόμη και σήμερα, παρά το ότι δεν είναι η κανονική διαδικασία, επιτρέπουμε στον κύριο Υπουργό να εκφραστεί επ' αυτή τη ε, έκθεση και συγκεκριμένα του σχεδίου έκθεση γιατί είναι ακόμη σχέδιο. Και θα δούμε πώ θα διαμορφωθεί κατόπιν. Η έκθεση αυτή, να το διευκρινίσω και αυτό, δεν είναι πρόσκληση διαπραγματεύσεων με την Ουγγρική κυβέρνηση. Η έκθεση αυτή θα σταλεί στο Συμβούλιο και καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει εάν θα ξεκινήσει μια διαδικασία κατά ενός κράτους μέλους εφόσον θεωρήσει ότι απομακρύνεται από το, τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αρχικά, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ανέφερε διάφορα θέματα που θα έπρεπε να απασχολήσουν τη ΛΥΜΠΕ. Ήταν μακροσκελής αυτός ο κατάλογος. Όλα τα θέματα αυτά τα εξέτασα, αλλά τα συγκέντρωσα σε ορισμένα θέματα. Ξεκίνησα με θέματα συνταγματικά, δικαστικά, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία της πανεπιστημιακής κοινότητας και ελευθερία θρησκείας. Και αυτό το έκανα γιατί ήθελα να καταλάβει και η κοινή γνώμη στην Ουγγαρία τι προβλήματα δημιουργούνται. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες αρμόζουν προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και πρέπει όλοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον νόμο. Εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες μεταξύ ημών και οι, οι Ούγγροι πολίτες πρέπει να θεωρούμε ότι μα σέβονται και μα προστατεύουν και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε το καθήκον. Εάν μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση να δεν ε, προστατεύει αυτά τα δικαιώματα, να παίξουμε το ρόλο μας. Πριν από δύο εβδομάδες παρουσίασα για πρώτη φορά την έκθεση. Και, όπως ήδη εξήγησα και θεωρώ σημαντικό να εξηγήσω και σήμερα, όλα όσα σημειώνω βασίζονται σε εκθέσεις από σώματα που ε, είναι ιδιαίτερα ε, αξιόπιστα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη. μελέτη επίση και αποφάσει των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου. Και είναι ιδιαίτερα εύγλωτο το γεγονό ότι έχουν γραφτεί τόσο πολλέ εκθέσει για τα θέματα τη Ουγγαρία τα περασμένα χρόνια. Επειδή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να βασιστεί αυτή η έκθεση σε στοιχεία και να ελέγξω και να ξαναελέγξω το περιεχόμενο αυτή τη έκθεση. Η έκθεση που έχετε ενώπιον σα έχει ημερομηνία 12 Απριλίου. κατάφερα να συμπεραλάβω, να συμπεριλάβω και ε, τα προκαταρκτικά πορίσματα του ΟΑΣΕ στην έκθεσή μου. Πορίσματα από τις ε, Ουγγρικές εκλογές. Και θα επιχειρήσω, εάν φτάσουν έγκαιρα, να συμπεριλάβω και τα τελικά πορίσματα του ΟΑΣΕ. Φυσικά, η έκθεση πρέπει να ενημερωθεί για να συμπεριλάβει και ονότα που είναι εξέλιξη. Και ιδιαίτερα να λάβει υπόψη αυτά που προσπαθεί να κάνει η Ουγγρική κυβέρνηση με το λεγόμενο νόμο «Σταματήστε το Σόρος». Όχι στο Σόρος. Βεβαίω εξετάζω πολύ περισσότερα θέματα ευρύτερα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου. Λαμβάνει υπόψη και παραβιάσεις σε θέματα αρμοδιότητας ε, αποκλειστικής ενός κράτους μέλους. Επίσης, περιλαμβάνει θέματα που έχουν ε, κοινωνικές επιπτώσεις και που δεν ε, αποτελούν ή δεν αποτελούν ακόμη παραβιάσεις του νόμου. Αλλά ε, είναι γεγονότα και που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ότι το κράτος δίνει το διαφημιστικό του υλικό μόνο σε κάποιες εφημερίδες ή ανακληθήσα νομοθεσία που ακόμη έχει αποτελέσματα, όπως ε, η ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών ή διάφορα θέματα που αφορούν διαδικασίες επί παραβάση, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε όχι. Δεν είναι μόνο ο γραπτός νόμος. Είναι και οι επιπτώσεις που έχει ο νόμος. Είναι τα οδυνηρά αποτελέσματα που έχουν κάποια νομοθετήματα στην κοινωνία. Καταλήγοντας. Νομίζω ότι κάναμε μια δουλειά ιδιαίτερα μεθοδική και πλήρη. Και κατέληξα ότι η Ολομέλη είχε δίκιο όταν είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία αποτελεί σαφή κίνδυνο σοβαρή παραβίαση των αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ένωση. Σημειώνω ότι τέσσερι επιτροπέ του σώματο έδωσαν γνωμοδοτήσει, οι δύο έχουν ήδη ψηφιστεί, η ΑΦΚΟ πριν από δύο εβδομάδε και η ΚΟΝΤ χθε ενέκριναν τις γνωμοδοτήσει του και οι δύο επιτροπές μας καλούν εμά ως ΛΥΜΠΕ όντω να προχωρήσουμε για να προσπαθήσουμε να πυροδοτήσουμε μια διαδικασία άρθρου 7.1. Στηρίζουν δηλαδή τη δουλειά μας. Καλό τους συνάδελφους να κάνουν σχόλια για να διευρύνουν και να βελτιώσουν την έκθεσή μου. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι σκιώδεις. Καταλαβαίνω ότι όλοι θα θέλετε το λόγο, όλοι οι παρόντες, οπότε σας παρακαλώ όλοι και οι σκιώδεις να μιλήσουν μόνο δύο λεπτά. Εάν δεν υπάρξει σφιχτή διαδικασία θα υπερβούμε το όριο της μίας ώρας. Θέλετε πάρα από δύο λεπτά. Ωραία. Ωραία. Τρία λεπτά για τους σκιώδες. Αλλά όλοι οι άλλοι δύο λεπτά. Η κυρία Σαζοντίνη σας έδωσε πολύ καλό παράδειγμα. Της έδωσα δέκα, πήρε έξι. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε. Τρία λεπτά οι σκιώδες. δύο υπόλοιποι. Πρώτος ο σκιώδης του ΕΛΚ. Η Ρομπέρτα Μετσόλα. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η έκθεση για την κατάσταση στην Ουγγαρία είναι άνευ προηγουμένου. Δυστυχώ έτσι έχει κατάσταση στην Ένωση. Ευχαριστώ την συγκίτρια για την προσέγγιση τη. Κάναμε πολλέ συνεδριάσει των σκιωδών. Έχω συμμετάσχει σε σχεδόν όλε. Ο στόχο ήταν να είναι μια τεκμηριωμένη και σύντομη παρουσίαση τη κατάσταση τη Ουγγαρία. Και είχαμε και την ε, συνάντηση με τον πρέσβη που ήταν και αυτή πολύ χρήσιμη. Να θέσω μερικά ερωτήματα. Ελπίζω να απαντηθούν. Ακούσαμε ότι στην Ουγγαρία η ελευθερία της πανεπιστημιακής κοινότητας, η ελεύθερη έκφραση και η, η, η δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων θίγονται και δίθηκε, δόθηκε το παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης. Δόθηκε μια περαιτέρω προθεσμία στα ξένα πανεπιστήμια για να ε, συμμορφωθούν με κάποιε προποθέσει, αλλά λέγεται ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα για τη δημιουργία βεβαιότητα για τον τρόπο λειτουργία των πανεπιστημίων. Ποιο θα θελήσει να, γίνει, να υποβάλει αίτηση για να γίνει φοιτητή στο πανεπιστήμιο, αν δεν ξέρει αν θα λειτουργεί το πανεπιστήμιο όταν θα αρχίσει η ακαδημαϊκή χρονιά. Καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν έχει προσφύγει κατά τη Ουγγαρία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αυτό. Υπάρχει θέμα διαφάνεια των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Ο Σκιώδης, όχι ο συντονιστής ε, του ΕΛΚ. Νομίζω ότι το νομοθέτημα αυτό προσπαθεί να περιορίσει τη δραστηριότητα αυτών που αποκαλούνται ξένοι πράκτορες. Όλοι θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογοι και ε, ε, άσκοποι παρέμβαση στη δυνατότητα της ελευθερίας ε, έκφρασης και του συνεταιρίζεστε. Γιατί πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση να παραβιάζει θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Καμία εκλογική πλειοψηφία δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά τα δικαιώματα. Αργότερα θα ρωτήσω και τον Υπουργό. Καλωσορίζω βεβαίως την παρουσία του. Εκτιμώ οποιοδήποτε είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει σε ένα διάλογο για να προκύψει μια λύση με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, όπω είδαμε και στη χώρα μου, τη Μάλτα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι υπουργοί έρχονται εδώ και την επομένη όταν γυρνάνε στο, στην ε, χώρα τους αρχίζουν ε, εκστρατείες κατά των Βρυξελών και μάλιστα και εμένα προσωπικά μου έχουν επιτεθεί. Ξέρω τι κάνει αυτή η κυβέρνηση στην Ουγγαρία. Τέλος. Ανησυχούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι η Ουγγαρία παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων. Γιατί ε, θεωρούμε ότι είναι λυδία λήθους. ο τρόπος αντιμετώπισης των προσφύγων για το πόσο λειτουργεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και πόσο ευρωπαίοι είμαστε. Ε, προσλέπω λοιπόν στην περαιτέρω εργασία το θέμα αυτό. Ξέρω ότι πολλά μέλη της πολιτικής μου ομάδας θα υποβάλουν πολλές τροπολογίες για όλα τα θέματα που αναφέρει η έκθεση και θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε ακριβώς στις ανησυχίες που εκφράζουν πολλοί για πολλά θέματα στη χώρα. Ευχαριστώ. Σκιώδης των Σοσιαλιστών, ο Ιώζε Δύο λεπτά. Ελπίζω να μου φτάσει ο χρόνος. Γιατί πρέπει να κάνω μερικές ε, θεμελιώδεις παρατηρήσεις. Μας απασχολεί από το 2012, εδώ και έξι μακριά χρόνια η κατάσταση στην Ουγγαρία. Για να δούμε εάν και κατά πόσο ανταποκρίνεται η κατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Ουγγαρία, αυτά που λέει το άρθρο 2 λοιπόν. Δεν συμφωνούμε όμως τι επιπτώσεις θα πρέπει να έχει αυτή. Για παράδειγμα, η διαδικασία του άρθρου 7 θα πρέπει να είναι μόνο ίστατη προσφυγή. Πρέπει να επιδιώξουμε πρώτα πολιτικές ε, λύσεις και να υπάρχει ένα όργανο όπως προτείναμε για μια τέτοια πολιτική αντιμετώπιση σε χαμηλότερο επίπεδο δεν έχει ακόμη γίνει δεκτή. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε όμως τα προβλήματα, γιατί δεν επιλύονται από μόνα τους. Διότι δυστυχώς έχει αναπτυχθεί μια παράλληλη πραγματικότητα στην Ουγγαρία, η οποία έχει τεκμηριωθεί, έχει κατοχυρωθεί, συγγνώμη, και μπορεί να αποτελέσει απειλή κατά της Φιλελεύθερης δημοκρατίας που είναι η έδρα της ε, Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει όμως, για να καταστεί σαφές, δεν υπάρχει μη φιλελεύθερη δημοκρατία. Διότι η φιλελεύθερη δημοκρατία βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση, στο δεχοσμό των ε, εξουσιών και σε μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Και πρέπει να σας πω, γιατί δεκαετίες ε, η Ανατολική Ευρώπη είχε τέτοιου τύπου εμπειρίες. Τότε λεγόντουσαν λαϊκές δημοκρατίες και ήταν τραγικές οι επιπτώσεις τους. Οι αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως τις ε, περιέγραψα, είναι αναγκαίε. Αλλιώ είναι κενή περιεχομένου η δημοκρατία αυτή. Είναι σαν κενό κτίριο. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίω η λειτουργία τη δημοκρατία ε, έχει ω στόχο να διαμορφωθούν πλειοψηφίε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με δημοκρατικό, με αντικειμενική πληροφόρηση. Οι τελευταίες εκλογές στην Ουγγαρία είχαν καθαρό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό και οι αμφιβολίες που εκφράστηκαν για το αποτέλεσμα, για αυτές τις εκλογές πρέπει να διευκρινιστούν συντόμως. Αλλά δεν είναι το βασικό μας θέμα, είναι μάλλον περιφερειακό. Το κεντρικό ερώτημα είναι τι δικαιώματα έχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Και συμφωνώ με τη σκιώδη του ΕΛΚ. Το θέμα είναι ποια είναι τα όρια οποιασδήποτε πλειοψηφία. Γιατί η δημοκρατία σημαίνει πάντα προστασία και των μειονοτήτων και των μειοψηφιών. Για να μπορεί να υπάρχει σωστή δημοκρατική ζωή. Περί αυτού πρόκειται. Δεν θέλουμε να κάνουμε καμία πολιτική κρίση για το πώς λειτουργεί η Ουγγαρία. Αυτό είναι θέμα του λαού της Ουγγαρίας. Γι' αυτό επιλέξαμε μία μέθοδο που μας επέτρεψε, επέτρεψε με σύνεση και ηρεμία να αποτιμήσουμε την κατάσταση της Ουγγαρίας και θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που απέφυγε τις ε, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και είναι λυπηρό που δεν υπήρξε πλειοψηφία για να στείλουμε μία αποστολή για να διαρευνήσουμε την κατάσταση στην Ουγγαρία. Η Επιτροπή της Βενετίας και η ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, όμως έκανε τέτοιες αποστολές και χαίρομαι που έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα των αποστολών αυτών η συγγήτρια. Είναι σαφής η έκθεση, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι στην περίπτωση της Ουγγαρίας έχουμε συστηματική παραβίαση του άρθρου 2, 2 των αρχών που περιέχει. Παρουσίασα την έκθεση αυτή στην ομάδα μου, υπήρξε ομόφωνη στήριξη και φυσικά θα υποβάλουμε και τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλουμε εγκαίως. Η Μαρία Κτζούρικ τώρα. Ο Μαρία Κτζούρικ, συγγνώμη, από Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν διάβασα το σχέδιο αυτό έκθεσης, σκεφτόμουν τον Winston Churchill. Αυτός ήρθε στο μυαλό μου. Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει μια γνωστή αλήθεια ότι δηλαδή η κοινοβουλευτική δημοκρατία με όλα τις τα πλεονεκτήματα πρέπει να δίνει μάχη κατά των μειονεκτημάτων της συνεχώς. Και εδώ έχουμε μια παρήθμιση φαινομένων που είναι παρόντα σε κάθε δημοκρατική χώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ειδικά την Ουγγαρία κατηγορούμε τώρα. Έχουμε τρία λεφτά μόνο στη διάθεσή μας, οπότε θα σας πω λίγα. Το θέμα της ένταξης των Ρώμα είναι ένα φαινόμενο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και για άγνωστο λόγο, μόνο η Ουγγαρία κατηγορείται ότι η ένταξη αυτή δεν γίνεται ικανοποιητικά, παρόλο που κάνει περισσότερα από άλλες χώρες. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι και τόσα πολιτικά κόμματα ε, ακολουθούν τις προκαταλήψεις τους ε, τελικά. Όπως και η κυρία Γέροκα, η αντιπρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου, που είπε τι κάνει η Ουγγαρία προκειμένου να εντάξει τους Ρωμά εκεί. Πώς είναι δυνατόν να αγνοούμε λοιπόν την πραγματικότητα εδώ μέσα. Στην ομάδα εργασίας μας, ο καθηγητής Γκάμπορ Πάλκιοκ από το Πανεπιστήμιο του Πίλτς, όταν απάντησε στις ερωτήσεις μου, παραδέχτηκε ότι οι κατηγορίες σε βάρος της Ουγγαρίας θα μπορούσαν να ισχύουν κάλλιστα και για τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του προηγούμενου Πρωθυπουργού. Όμως τότε κανένας δεν ανησύχησε για το πώς λειτουργεί το κράτος, τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Οπότε, περί πρόκειται τελικά. Πρόκειται για δημοκρατικές προδιαγραφές, αρχές. Η κυρία Χετφέλτ απάντησε ωραία σε αυτό το Δεκέμβριο που συναντηθήκαμε και είπε τότε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το νόμο της Ουγγαρίας με το κράτος δικαίου σε άλλες χώρες. Πολύ καλά, δηλαδή πρόκειται για επιλεκτική δικαιοσύνη εδώ που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή μεταχειριζόμαστε μια χώρα διαφορετικά από ό,τι μεταχειριζόμαστε τις άλλες. Σωστά το είπε λοιπόν και το επανέλαβε και στην Ολομέλεια. Υπάρχουν άνθρωποι ε, στους οποίους δεν αρέσει καθόλου η Ουγγαρία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να το συνειδητοποιήσουμε ότι περί αυτού πρόκειται. Και δεν πρέπει αυτό να διχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προλαλή σα είπε ότι δεν είναι η πλειοψηφία η οποία πρέπει δικτατορικά να επιβάλλει την απόψή τη στη μειονότητα. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, κοιταχτείτε στον καθρέφτη όλοι και πείτε μπροστά στον καθρέφτη σας ότι η πλειοψηφία δεν μπορεί δικτατορικά να επιβάλλει την άποψή τη στη μειονότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Λουί είναι ο επόμενος συντονιστής Α, όχι. Έχει αντικατασταθεί από την Νάταλη Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, ο Λουί Μισέλ δεν μπορούσε να είναι εδώ τώρα. Οπότε, εκ μέρους της ομάδας μας, της Άλτε, θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό το οποίο μας έχει μαζέψει εδώ σήμερα είναι η εξέταση μιας ιδιαίτερης έκθεσης. Μια έκθεση η οποία βέβαια μας θεσμεύει ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Εδώ πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες. Οι Ούγγροι αυτό ακριβώς είναι, Ευρωπαίοι πολίτες. Οπότε δεν κάνουμε καθόλου ε, δικηπροθέσεων σε βάρος των Ούγγρων. Κάθε άλλο. Πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει με τη συνέπεια, με τη συνοχή του συνόλου, με αυτό το οποίο μας ενώνει όλους και αυτό το οποίο μας ενώνει είναι η αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Μεταξύ αυτών και των Ούγγρων βεβαίως. Οπότε, ευχαριστώ βέβαια την Τσούντιθ Σατζετίνη, την εισηγήτριά μας, για την τόσο καλή δουλειά που έκανε, τη λεπτομερή που μας επέτρεψε να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη έκθεση, μετρημένη, ε, συνεκτική, η οποία επιβεβαιώνει τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων απέναντι στις συνθήκες. Βασίζεται η έκθεση αυτή σε αναλύσεις που έχουν γίνει από διάφορους διεθνείς οργανισμούς πλουραλιστικούς, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και ο λόγος τους μετράει γιατί είναι αξιόπιστοι. Και μαζί με τον Λουί Μισελ λοιπόν που είναι σκιώδης συγητή, συμφωνούμε με την άποψη και την προσέγγιση της συγητρίας όσον αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά τον κατακαιρματισμό της δικαιοσύνης και όσον αφορά το σεβασμό της δημοκρατίας, των μειονοτήτων, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτησία δικαιοσύνης κλπ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν και προσοχή περιμένουμε την απάντηση του Συμβουλίου. Η Σόφιν Χετβέλτ ε, αναφέρθηκε από τον συνάδελφο του ECR, θα απαντήσει ε, βεβαίως ε, σε αυτά τα fake news θα έλεγα εγώ που ανέφερε ο συνάδελφος που ουσιαστικά μεταφέρει λάθος τα λόγια της συναδέλφου. Τα παραμορφώνει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Γκουέντζιαρ. Η Μαρή Κριστίν Βερζιά είναι η σκιώδη συζητήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντως είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η στιγμή που ζούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη έκθεση αυτού του είδους που κάνουμε και η κυρία Σορτζεντίνη είχε μπροστά της μια πραγματική πρόκληση. Νομίζω όμως ότι τα κατάφερε. αναφέρθηκαν προκαταλήψεις, πολιτικές προκαταλήψεις, δίκη προθέσεων. Στην έκθεση αυτή όμως η κυρία Σαρτζεντίνη επέλεξε να βασιστεί σε αποφάσεις διεθνών οργανισμών αναγνωρισμένων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την ευχαριστώ που ακολούθησε αυτή την οδό. Θα σταθώ σε κάποια σημεία που πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Το θέμα πρώτα απ' όλα της προστασίας δεδομένων. Βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην απόφαση της ότι είναι πολύ καλό αυτό που έκανε. Έπειτα το θέμα της ελευθερίας έκφρασης. Πολύ σωστά μετά την αποστολή παρατήρησης των εκλογών της ΟΑΣΕ βασίστηκε και στον ΟΙΕ για αυτά. Το θέμα της ελευθερίας της θρησκευτική, που σημαίνει ότι πρέπει κανείς να έχει το δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει σε κάτι. Το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων, σε αυτό θα επανέλθω ε, όταν θα μιλήσω για το πακέτο σε βάρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έπειτα φύγει το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Βασίζεται στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων και νομίζω ότι όλα αυτά πολύ καλά αποτελούν τη βάση ε, του κειμένου, γιατί έχει να κάνει και με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και σε αυτό θα επανέλθω στη συνέχεια. Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη διαφθορά και στη σύγκρουση συμφερόντων, δεν αναφέρεται η Όλαφ. Παρ' όλα αυτά, η Όλαφ έχει θίξει το θέμα και η δικιά μας Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών έχει αναφερθεί σε αυτό. Η Όλαφ λοιπόν έχει κάνει πολλές έρευνες και συστάσεις που αναφέρονται ακριβώς σε παρατυπίες, σε σύγκρουση συμφερόντων και σε κακή οργάνωση. Θεωρεί η Όλαφ ότι θα έπρεπε να επιστραφούν πολλά εκατομμύρια ευρώ από την Ουγγαρία οι συστάσεις της βασίζεται σε στοιχεία από τις εθνικές αρχές. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί η Ουγγαρία αντιτίθεται στο, στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και γιατί δεν, μπορεί να, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα προκειμένου να υλοποιήσει τις συστάσεις της Όλαφ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δικιά του έκθεση δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το θέμα. Έρχομαι τώρα στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Εδώ θέλω να μιλήσω για το πακέτο αυτό κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όχι για το όχι στο σώρος, το οποίο είναι μια γνωστή υπόθεση. Εμένα με απασχολεί η απουσία δικαστικών μέσων. Στην περίπτωση που μία οργάνωση δεν έχει δικαίωμα πια να δρά εδώ είναι το θέμα της ελευθερίας συνεταιρίζεστε. Ακόμα και ευρωπαϊκά κονδύλια δεν μπορούν να δοθούν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Πετύχαμε βέβαια μετά τις ε, εκλογές να το ξαναδεί αυτό το θέμα η κυβέρνηση. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αντί τελικά να επιταχύνεται η διαδικασία διόρθωσης, καθυστερεί. Και θα έλεγα εγώ ότι αν δεν έχουμε νέα στοιχεία πολύ γρήγορα, περιμένουμε αρχές Ιουνίου την ε, νέα άποψη της Επιτροπής της Βενετίας. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να σταθεί σε αυτά. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία λοιπόν για να καταλήξουμε στο ότι υπάρχει συστηματική, για να μην πω και συστημική παραβίαση των θεμελιωδών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπω παραγράφονται στο άρθρο 2 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσα, Πρόεδρε. Ο κίνδυνο είναι ότι Έχουμε πολλά μέλη που θα θέλουν να μιλήσουν και μετά την παρέμβαση του Υπουργού και ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Τέλος πάντων το λέω αυτό. Η κυρία Φεράρα για το FDD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Σερτζεντίνη, για την εξαιρετική δουλειά και για την ε, εις βάθος έκθεση. Εγώ Ήμουν εισηγήτρια για την κατάσταση του σεβασμού των ευρωπαϊκών των δικαιωμάτων στην Ευρώπη για το 2013-2014 και τότε μιλούσαμε για την αναγκαιότητα παρακολούθησης χώρα για να εγγυηθούμε το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να προλάβουμε την παραβίασή τους ήδη. Ε, τότε ε, υπήρχαν κάποιοι φόβοι ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα είδος ε, μαύρου καταλόγου για τις κακές χώρες όπως αποκαλούνταν. Και η ανησυχία ήταν ότι θα μπορούσαμε να θίξουμε ευαισθησίες κάποιων χωρών όπως η Ουγγαρία που ήταν τότε στο στόχαστρο για αφαιρόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βέβαια, αν ε, δεν θέλουμε να είναι υποκριτική η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το σεβασμό των κριτηρίων της ε, Κοπενχάγης ε, πριν την ένταξη και κατόπιν αφού μπει αυτή η χώρα τα ξεχνάμε όλα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε πώς έχει η κατάσταση σε σχέση με το σεβασμό των θελημένων δικαιωμάτων σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εγγυόμαστε ότι κάθε χώρα τη στιγμή που αποφασίσει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται τις ε, αρχές τις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το κράτο δικαίου. Επομένως ε, δεν ε, θέλουμε μια Ευρώπη à la carte και να αποφασίζει κάθε κράτος μέλος τι το βολεύει και τι δεν το βολεύει. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνε του απέναντι σε ευρωπαϊκά αν όχι παγκοσμία φαινόμενα. Τώρα θέλω να αναφέρω ε, μια συγκεκριμένη απόφαση, ε, μια συγκεκριμένη υπόθεση έχει να κάνει με το ε, διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Από ό,τι φαίνεται η Ουγγρική κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της στον τομέα αυτό. Μάλιστα φαίνεται ότι αρνείται να δεχτεί την μετακατάσταση των προσφύγων. Μάλιστα, μιλάμε και για παράνομη κράτηση ανηλίκων καθ' όλη την διαδικασία. Ε, από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποφεληθεί και από τα κονδύλια που έρχονται από τις Βρυξέλλες, Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ε, πέρα από τα ωφέλη υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις για τα κρατη Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να σέβεται κανεί ε, είναι το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπρίμηση, εγώ θα ήθελα να υπάρχει η βούληση, να υπάρχει μια προσεκτική παρακολούθηση και τη Ουγγαρία αλλά και των υπολείπων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά τη Ουγγαρία θα ήθελα να υπάρχει βούληση στο να συνεργαστεί γιατί την, ε, να μα εγγυθεί ότι σέβεται το κράτο δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που σεβαστήκατε και το χρόνο. Να πάμε τώρα στον ε, κύριο Σιάρτο. Η συγγήτρια έχει συμφωνήσει για την παρουσία του εδώ και μπορεί να τοποθετηθεί για την έκθεση. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργό για 10 λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για την πρόσκληση στη σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη απόφαση να ε, επιτρέψετε ε, στο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τον εγκρικό λαό να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα κατά τη ε, εκφώνηση των εισαγωγικών μου παρατηρήσεων αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Καταρχήν να σας ενημερώσω για το τι συνέβη πριν μισή εβδομάδες. Είχαμε κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία και ε, υπήρξαν ε, από εξωτερικούς παράγοντες που προσπάθησαν να αποδυναμώσουν τη θέση της Ουγγρικής κυβέρνησης. Και σε αυτό τον οίκο υπήρξαν πολλοί που προσπάθησαν να επηρεάσουν ε, το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία. Και μάλιστα σε αυτή την πόλη ε, υπήρξαν ε, κάποιες πληροφορίες που διαδόθηκαν για να βοηθηθεί η Ουγγρική αντιπολίτευση. Ίσως θα πρέπει λοιπόν από κοινού να αξιολογήσουμε, να εξετάσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Είχαμε συμμετοχή ε, στις εκλογές της τάξης του 70%, πολύ ψηλή συμμετοχή, 49,6% των ε, ψήφων ε, ήταν υπέρ του Φιντές. Το Φιντές έλαβε 2 εκατομμύρια 800.000 ψήφους και ουσιαστικά είχαμε σχεδόν ένα εκατομμύριο ψήφους παραπάνω από το δεύτερο κόμμα οι Ούγγροι που θέλετε να τους προστατεύσετε, που δεν ξέρω από ποιον, μίλησαν ξεκάθαρα για τα τελευταία οκτώ χρόνια, ε, έδωσαν την αξιολόγησή τους, έκαναν την αξιολόγησή τους και μάλιστα δήλωσαν ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν τα επόμενα έτη. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη και να σαβαστείτε τις δημοκρατικές αποφάσεις των Ούγγρων, να μην τις αμφισβητείτε, ούτε να τιμωρείτε τη βούληση αυτών. Βέβαια, μπορεί να μην συμφωνείτε με την απόφαση των Ούγγρων, μπορεί να σας δημιουργεί σύγχυση το πώς αποφάσισαν οι Ούγγροι πριν δυόμιση εβδομάδες, όμως οι Ουγγροί μπορούν να λάβουν μια απόφαση για το μέλλον της Ουγγαρίας, ενώ εσείς δεν είστε στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορείτε να λάβετε τέτοιες αποφάσεις. Πριν δύο μισή εβδομάδες υπήρξε μια ξεκάθαρη επιλογή ενώπιον του Ουγγρικού λαού, γιατί προσφερόταν ε, μια προσφορά αντιμεταναστευτική για την προστασία των Ούγγρων θα μπορούσε να γίνει μια άλλη επιλογή που προτινόταν από τη ΣΜΚΙΟ και την αντιπολίτευση. Όμως έγινε η επιλογή από τους Ούγγρους και μας αναθέτει ένα ξεκάθαρο καθήκον ότι η Ουγγαρία δεν θα είναι μια χώρα υποδοχής μεταναστών. Έτσι λοιπόν είμαι έτοιμος να συνεχίσω την έντονη συζήτηση για το μεταναστευτικό με την Επιτροπή σα, όμω είμαστε έτοιμοι, γιατί εμεί θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε την πορεία μα και πιστεύουμε ότι μόνο οι Ούγγροι πολίτε μπορούν να αποφασίσουν για το ποιο επιτρέπεται να μπει στη χώρα και με ποιον θέλουν να ζήσουν στην ίδια του τη χώρα. Εμεί θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας, προστατεύοντας ε, την ασφάλεια των πολιτών και της χώρας μας. Δεν θα δεκτούμε υποχρεωτικές ποσοστώσεις ούτε θα δεκτούμε ότι μια πιο πολυπολιτισμική κοινωνία είναι πιο πολύτιμη από μια ομοιόμορφη κοινωνία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους Ούγκρους και την Ουγγαρία. Έχουμε τώρα μία συλλογή κατάφορων ψεμάτων στην εισηγήτρια μαγείρευσε την έκθεση αυτή, έλαβε υπόψη της σε διάφορα, αλλά όχι τα γεγονότα. Λέτε ότι δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων ενημέρωση στην Ουγγαρία. Αυτό είναι ψέμα. Τα μέσα ενημέρωσης ε, είναι πολύ περισσότερα και διαφοροποιημένα στην Ουγγαρία δεν μπορείς το χάρη στην Ουγγαρία να κρατήσεις ε, κρυφό ότι ε, παράνομοι μετανάστες διαπράττουν εγκλήματα στην Ουγγαρία κατά των πολιτών. Αυτό δεν αποκρύπτεται από τα μέσα μεζικής ενημέρωσης Στην Ουγγαρία ε, υπάρχουν ε, ε, ισότιμα στον αριθμό, εισάριθμα, συγγνώμη, ε, τηλεοπτικά κανάλια που είναι δημόσια όπως και ιδιωτικά της αντιπολίτευσης. Υπάρχει πολύ σημαντική κριτική που ασκείται κατά της Ουγγρικής κυβέρνησης και αν δείτε τις διάφορες ιστοσελίδες, ε, πολλές επικρίνουν την ε, Ουγγρική κυβέρνηση. Τώρα, στην εκλογική εκστρατεία. Στην προεκλογική εκστρατεία υπήρξαν ε, κάποια έγγραφα που διαδίδηκαν από τις Βρυξέλλες και εκεί περιλαμβάνονταν ψέματα και κατηγορίες ε, κατά κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Και την ημέρα των εκλογών ε, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, γιόρτασαν την υψηλή συμμετοχή γιατί πίστεψαν ότι θα οδηγήσει σε ήττα ε, του κυβερνώντος κόμματος. Όμως ε, δεν ήταν έτσι. Η έκθεση ε, λέει ότι οι ΜΚΟ καταπιέζονται στην Ουγγαρία. Έχουμε 65.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ουγγαρία. Κάποιες πράγματι παραπονιούνται, αλλά μόνο αυτές που έχουν καταστεί ανοιχτοί πολιτικοί παίκτε που συμμετείχαν στην προεκλογική εκστρατεία και προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν του ανθρώπου να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αυτές ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν λάβει σημαντική χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι οι Ούγγροι έχουν το δικαίωμα να ξέρουν αν ε, αυτές οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό, ε, ποιον εκπροσωπούν, τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζουν. Αυτές οι ΜΚΟ πάντοτε ζητούν διαφάνεια. Αν είστε υπέρ τη διαφάνειας, ε, γιατί δεν λέτε από πού παίρνετε τα κονδύλια. Αν ε, ντρέπονται να το αποκαλύψουν, ε, τότε εμείς δεν μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι ότι στην έκθεση τολμάτε και αναφέρετε ότι αποτελεί πρόβλημα ο αντισημιτισμός στην Ουγγαρία. Κοιτάξτε, αυτό το απορρίπτω κάθετα. Γιατί Καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει τόσο πολλά κατά τον αντισημιτισμού όσο η Ουγγαρία. Γιατί ε, ουσιαστικά ε, βλέπουμε κάποιες ε, επιθέσεις να γίνονται κατά των Εβραίων σε άλλες χώρες, ενώ στην Ουγγαρία έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα Εβραίων και χρησιμοποιούνται ουγγρικά κονδύλια και το 2000 ε, ε, μπορώ να σας πω και ότι η άρνηση του λοκαυκώματος είναι πάρα πολύ σοβαρό δίκημα στον ποινικό μας κώδικα. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι ορισμένα ξεκάθαρα παραδείγματα για το ποιο είδους γεγονότα βάζετε σε αυτή την έκθεση και ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο μηχανισμός ε, που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη της ε, έκθεσης ε, αυτής. Είστε ε, ουσιαστικά μεροληπτικοί απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική και ασκείτε κριτική στην Ουγγαρία ε, για το τι κάνει στον τομέα αυτό, εσείς ε, και επειδή δεν μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή την ε, φιλομεταναστευτική σας ε, πολιτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τη βούληση του γκρικού λαού δεν θα σας επιτρέψουμε να εφαρμόσετε το σχέδιο Σόρος, το σχέδιο μετανάστευσης στην Ουγγαρία. Και θα προστατεύσουμε όχι μόνο την Ουγγαρία, αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σας ευχαριστώ που με καλέσετε για να σας πω την αλήθεια για την Ουγγαρία. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, όσοι δεν είναι μέλη τη Επιτροπή μας, ε, να μην χειροκροτούν. Πρέπει να έχουμε κάποια πειθαρχία και κάποια αξιοπρέπειες διαδικασίε μα. Λοιπόν, εννέα συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Ε, αυστηρά με τη σειρά με την οποία ε, δήλωσαν ε, το αίτημά του στη γραμματεία. Σας παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Η εισηγήτρια επέτρεψε στον Υπουργό να λάβει το λόγο, είχε συμφωνηθεί και συμφωνήθηκαν και οι χρόνοι. Η εισηγήτρια θα ολοκληρώσει το τέλος, θα κάνει το κλείσιμο. Και τώρα θα πάρουν τα, το λόγο οι συνάδελφοι. Θα διαβάσω το κατάλογο και θα τον κλείσω. Με τη σειρά που ε, δήλωσα στη γραμματεία. Μίστερ Μπόνι, Μίστερ Μπέκερ, Becker, Γκάου, Μίστερ Αλμπρέχτ, Albrecht, Γιουρόκα, Mrs. Ιντεβέλτ, και Mrs. Κουτζίσκα. Είχατε ζητήσει κι εσείς. Συγγνώμη, έχουμε και δύο που δεν είναι μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Μόρβάη και η κυρία Ζ... και ο ο κύριος Βέρ, λοιπόν. Κλείνω ο Ο κύριος Νίντο Μίλο είναι πρώτος. Σας παρακαλώ ησυχία. Κύριε Νίντο Μίλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κάνατε μία αναλυτική παρουσίαση του τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε τι εκλογέ. Αλλά ξέρετε το θέμα μας εδώ δεν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Κανεί δεν αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών. Εγώ θέλω να ασχοληθώ μεταξύ τα τρία θέματα. Είπε ο κύριο Υπουργό ότι τα μέσα είναι ελεύθερα στην Ουγγαρία. Ότι υπάρχει πλήρη ελευθερία των μέσων. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση διεθνής έκθεση που τονίζει ότι η Ουγγαρία είναι στην 76η θέση του καταλόγου των χωρών από πλευράς ε, ελευθερίας των μέσων και έχει πέσει από την προηγούμενη θέση της που ήταν ψηλότερη και από το 2010 Επίσης έχει, βελτιωθεί, έχει συγγνώμη, επιδεινωθεί η κατάσταση όσον αφορά την διαφθορά στην Ουγγαρία. Και αυτό είναι πόρισμα της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, της οποίας η Πρόεδρος ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με εσάς, κύριε Υπουργέ. Κάτι γενικότερο. Η δημοκρατία ε, προϋποθέτει ότι δεν θεωρούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους ως εχθρούς. Η δημοκρατία παρέχει χώρο και προστασία σε όσους έχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν ε, συντάσσει καταλόγους και δεν παρακολουθεί όσους έχουν άλλες απόψεις. Η δημοκρατία δεν είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Είναι ο συνεχής αγώνας για συμβιβασμούς. Περί αυτού πρόκειται. Το θέμα δεν είναι αν θα καταδικάσουμε την Ουγγαρία ή την κυβέρνηση. Δεν είναι αν είναι κανείς υπέρ κατά της μετανάστευσης. Είναι εάν κανείς σέβεται τις βασικές αρχές της ε, Ουγγρικής Δημοκρατίας που θα πρέπει να σέβεται και η Ουγγρική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να μην χειροκροτείτε. Να μην χειροκροτεί κανείς. Μπόνι παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας καλέσαμε εδώ. Είστε προσκεκλισμένος μας και ο στόχος μας ήταν να έχουμε μια λογική και ήρεμη συζήτηση. Αλλά τελικά τι είδαμε. Εσείς ε, προτιμάτε να είστε πρωταγωνιστής αυτής της ε, αυταρχικής ε, στάσης. Κοιτάξτε πώς μιλάτε εσείς και πώς μιλάμε εμείς. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την θαυμάσια εργασία της που βασίζεται σε εκτεταμένη τεκμηρίωση. Το πακέτο κατά του όρους, σταματήστε τον όρους, είναι μια προσπάθεια να στιγματιστούν και να εκφοβιστούν άτομα και οργανώσεις. Θέλουν η κοινωνία των πολιτών να είναι υποχείριο της κυβέρνησης. Υπάρχουν αυθαίρετες και πολιτικά κινούμενες επιθέσεις κατά της ελευθερίας έκφρασης στην Ουγγαρία. Άλλη σοβαρή ανησυχία που αναφέρει η έκθεση. Συγκέντρωση των μέσων σε λίγα χέρια με σαφή στόχο επηρεασμού της κοινή γνώμης. Έχουν ε, καταλάβει όλους τους ραδιοσταθμούς και όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ορισμένη. Η Ουγγαρία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων αυταρχικών καθεστώτων. Η νομοθεσία κατά του σώρου ειναι είναι copy-paste της νομοθεσίας κατά τον ΜΚΟ που έχει εγκρίνει ο κύριος Πούτιν. Αυτό το αυταρχικό κύμα εκτιλήσεται και επεκτείνεται σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, το γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια τον κύριο Όρμπαν. Είναι πολύ λυπηρό να παρατηρώ ότι κατρακυλάει προς τον αυταρχισμό. Αλλά καταδεικνύει ότι η Ουγγαρία δεν είναι μεμονωμένο πρόβλημα. Ο αυταρχισμός ενισχύει τις απειλές κατά της δημοκρατίας σε ολόκληρη την Ένωση και περαιτέρω. Καλώ όλους τους συναδέλφους να μην αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να επαγρυπνούμε αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία μπορεί να συμβεί και αλλού. Εγώ είμαι Πολωνός. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στον ουγγρικό λαό ότι η ουγγρική κοινωνία των πολιτών δεν είναι μόνη. Δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο να κερδίσει κανείς εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέκα. Ευχαριστώ και εγώ χαιρετίζω το ότι εσείς είστε εδώ για να μας μιλήσετε. Ως ε, γείτονας, ως ε, φίλος, έχουμε το δικαίωμα να σας επικρίνουμε και να πούμε την ελευθερία. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Είναι πολύ ανησυχητικά ότι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Ουκρανίας, το Τζόμπικ, πήρε 20% των ψήφων με καθαρά ξενοφοβικά και καθαρά αντισημιτικά μηνύματα. Το Φιντές θα πρέπει να μη συμμετάσχει σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Να επιτίθενται σε άτομα για να αναφέρω από λόγους του Ουγγρού Πρωθυπουργού. Λένε, είμαστε κατά ενός εχθρού που είναι διαφορετικός από μας, που κρύβεται, που δεν είναι έντιμος αλλά πονηρός, που δεν είναι έντιμος αλλά ανέντιμος, που δεν είναι ε, εθνικός αλλά διεθνής, που δεν πιστεύει στην εργασία αλλά που είναι κερδοσκόπος, που δεν έχει πατρίδα αλλά κάνει σαν να ε, κατέχει ολόκληρο τον κόσμο το ψήφισμα του για τον αντισημιτισμό της Επιτροπής μας και που εγκρίθηκε με τρία τέταρτα από το σώμα μας από όλα τα πολιτικά κόμματα τέτοιες δηλώσεις που είναι ο ορισμός του αντισημιτισμού θα τις ε, δύο και ποινικό. Λέγεται ότι ο κύριος Όρμπαν ακόμη συνομιλεί με τον κύριο Σόρος αλλά αυτά που λέει είναι αντισημιτισμός. Και πολλοί Ούγγροι Εβραίοι, όχι μόνο στην Ουγγαρία βεβαίως, αλλά και στην Ουγγαρία είναι ε, ιδιαίτερα φοβισμένοι. Ως πρόεδρος ε, της διαπολιτικής ομάδας κατά του αντισημιτισμού πρέπει να καταδικάσω αυτές ε, τις δηλώσεις γιατί είναι υποκίνηση σε αντισημιτικές ενέργειες και καλό την Ουγγρική κυβέρνηση να σταματήσει αυτό το λεξιλόγιο και αυτές τις επιθέσεις. Όπου και αν συμβαίνουν αυτά βέβαια πρέπει να τα καταδικάζουμε. Σκεφτείτε το μέλλον των πολιτών στη χώρα σας. Το μέλλον τους ανήκει στην Ευρώπη. Δείξτε υπευθυνότητα. Για να αποφύγετε αυτές τις απειλητικές εξελίξεις. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή έκθεση. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή μα και για το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και αυτό το κάνει το σχέδιο έκθεση. Και δεν προσπαθεί να προκαλέσει ε, μικροπολιτικέ ε, διχογνωμίε. Αντίθετα, είναι θέμα θεμελιωδών αξιών τη Ένωση. σε όλα τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα το έχουμε σε πολλά κράτη-μέλη. Και αυτό είναι μια πρώτη αντιμετώπιση που θα αποτελέσει νομολογία. Πρέπει να δείξουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία, και το κράτος δικαίου είναι η βάση της ευρωπαϊκής πορείας. Και γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η Ουγγαρία έχει υπογράψει όλες αυτές τις συμβάσεις. Ισχύει λοιπόν το ενωσιακό δίκαιο και στην Ουγγαρία. Οι εκλεγμένοι λοιπόν στην Ουγγαρία δεσμεύονται από τις ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει υπογράψει ο λαός. Όσο είναι τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουγγαρία θα εξακολουθεί να ισχύει αυτό και θα πρέπει να τηρούν του κανόνε. Αυτό που είναι πολύ απογοητευτικό είναι ότι περίμενα θα συζητήσουμε επί του περιεχομένου με λογικό και έντιμο τρόπο. Αλλά αυτό που άκουσα είναι μία από τι πιο ξεδιάτροπε ομιλίε που έχω ακούσει ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρί κανένα σεβασμό. Και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Και ο τρόπο με τον οποίο ήρθατε εδώ για να μας κάνετε κηρύγματα προπαγάνδας. Δεν ασχολείστε καθόλου με τις επικρίσεις μας. Και γι' αυτό σας χειροκρότησε εδώ μόνο μία από το κόμμα σας στην Ουγγαρία. Και επιτρέπετε στον εαυτό σας να πείτε ότι δεν υπάρχει αντισημιτισμός στην Ουγγαρία. Κάθεστε δίπλα σε μία βουλευτή που είπε ότι οι Ούγγροι Εβραίοι. Παραθέτω ε, καλύτερα να παίξουν με το ε, όργανό τους το οποίο έχει υποστεί και περιτομή. Εκλέγεται στην Ουγγαρία το άτομο αυτό. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Πρέπει να αντιμετωπίσετε σοβαρά το θέμα αυτό. Γιατί όλα αυτά και αυτά είναι σαφής παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Ε, Γκάλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή είναι εξωφρενών. Δεν είναι αξιοπρεπής καθόλου. Το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να την κάνει. Οι παρεμβάσεις είναι πραγματικά αναξιοπρεπείς και δεν ταιριάζουν καθόλου στο κοινοβούλιο μας αλλά και στην Ουγγαρία και τους Ούγγρους πολίτες. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να φροντίσουμε να συμπεριφερόμαστε με εξωπρέπεια και αυτοί που μας προσβάλλουν θα πρέπει να ζητούν συγγνώμη στη συνέχεια. Δεν έχω χρόνο βέβαια να αναφερθώ σε όλα τα ψέματα και σε όλες τις τρευλώσεις, τις ε, δηλώσεις, τις λαθασμένες που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Όμως, παραθέτω από τα αγγλικά, ότι η κοινωνία δεν ε, παρακολουθεί τον νόμο. Αυτό είναι μια μεγάλη προσβολή για την Ουγγαρία και το Ουγγρικό έθνος. Πρόκειται για μια επίθεση στο κράτος δικαίου στην Ουγγαρία που ισχύει πάνω από χίλια χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσει συγγνώμη η συγκίτρια για αυτή τη δήλωση. Αλλά πάω και ακόμα πιο πέρα. Από αυτά που ακούω σήμερα, από αυτά που διαβάζω στην έκθεση αυτή, τις διάφορες σελίδες, γίνεται η περιγραφή μια χώρα σαν να επρόκειτο για μια δικτατορία στην Κεντρική Αφρική. Σαν να μην μιλάμε για μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έγιναν μάλιστα μόλι δημοκρατικέ εκλογέ. Υπάρχει ένα ε, καλώς λειτουργών ε, σύστημα ε, νομικό και είναι κάτι το οποίο αποτελεί προσβολή και για μένα προσωπικά αλλά και για ολόκληρο το ουκρικό λαό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξετε συμπεριφορά και ύφος λέτε ότι μιλάτε για γεγονότα, για στοιχεία, ενώ η έκθεση, η έκθεσή σας είναι, και οι δηλώσει σας είναι γεμάτες ψέματα, παραπλανητικά στοιχεία, όχι γεγονότα. Μιλάτε, λέτε, για το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ε, ΟΑΣΕ, τον ΟΙΕ κλπ. Και από πού παίρνουν τις πληροφορίες τους από τις ίδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τις ε, ίδιες οργανώσεις λοιπόν και τους ίδιους εμπειρογνώμονες. Δεν είναι αληθείς οι απόψεις αυτές και εσείς εκεί βασίζεστε σε αυτά τα ψέματα. Αρνούμε λοιπόν τις δηλώσεις σας. Δεν συνεργαζόμαστε με το Γιώμπικ που είναι το κόμμα της ακροδεξιάς. Αρνούμε τις κατηγορίες σας. Μας κατηγορείτε για πράγματα τα οποία δεν κάναμε. Αυτή είναι μια ψευδοδίκη. Εσείς έχετε εκ των προτέρων αποφασίσει για τις τύχες μας. Ακριβώς εξαιτίας της μεταναστευτικής μας πολιτικής και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Η κυρία Χετφέλτ. Ευχαριστώ πολύ. Πού να ξεκινήσω, πού να πρώτο ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα είναι μια κλασική περίπτωση αυτή ενός αυταρχικού καθεστώτος το οποίο έφτασε στην εξουσία με τον παραδοσιακό τρόπο που παριστάνει το θύμα, ότι άλλοι είναι οι εχθροί, υπάρχουν αντίπαλοι, υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον τους ε, που ψεύδεται. Είναι ένα παραδοσιακό παράδειγμα, κλασικό. Με εσείς δεν είσαστε κάποιος στον οποίο ανήκει ο Ουγγρικός λαός. Έχετε κλεγεί να εκπροσωπήσετε προσωρινά τον Ουγγρικό λαό. Και θέλω να το ξέρω γιατί άκουσα τα περισσότερα από αυτά που είπατε, μετά έβγαλα τα ακουστικά μου γιατί πραγματικά ήμουν έξαλλη και κουρασμένη από όλες αυτές τις κατηγορίες που μας απευθύνατε και τα ψέματα εναντίον μας. Με ποιο τρόπο πιστεύετε εσείς ότι εκπροσωπείτε το άλλο μισό του γκρικού λαού που δεν σας ψήφισε. Τις δεκάδες χιλιάδες ε, ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους κατά το αυταρχικού σας καθεστώτος. Αυτούς πώς τους εκπροσωπείτε νομίζετε. Αυτά που λέμε σήμερα δεν έχουν και τόσο σημασία γιατί είναι ξεκάθαρο ε, ότι υπάρχουν τα δικά σας μέσα ενημέρωσης που θα κάνουν προπαγάνδα και θα παρουσιάσουν όπως θέλουν τη σημερινή συζήτηση στον Ουγγρικό λαό. Εσείς θα είστε πάλι το θύμα και εμείς θα είμαστε οι εχθροί. Και άλλο εχθρό είναι ο κύριος Όρο, ο οποίο από ό,τι φαίνεται χρηματοδοτεί όλη αυτή τη συνωμοσία εναντίον σα. Μήπω θα πρέπει να ξέρουμε περισσότερο τα δικιά σας πηγή χρηματοδότησης... ...εκτός ε, του γεγονό ότι καταχράστε ευρωπαϊκά κονδύλια για του δικού σα διεφθαρμένου ηγέτε, μήπως από τον κύριο Πούτιν, μήπως από τον κύριο Πάντα, τον άλλον Αμερικανό που χρηματοδοτεί από ό,τι φαίνεται και του εταίρους του Πολωνικού Κόμματος. Μήπως λοιπόν, θα έπρεπε να κοιτάξουμε από πιο κοντά αυτή τη χρηματοδότηση. Και για να τελειώσω, Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πείτε μπράβο για την έκθεση, γιατί επιβεβαιώνει αυτά τα οποία θέλει να πετύχει ο κύριος Ορμπάν. Ένα διαφορετικό καθεστώς, ένα διαφορετικό σύστημα. Το είπε ότι θέλει να δημιουργήσει μία μη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αλλά υπάρχει, οπότε μάλλον για, αυταρχία, για αυτό, αυταρχικό καθεστώς εννοεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι ο κύριος Ορμπάν κάνει ακριβώς αυτό που θέλει, οπότε γιατί να διαφωνείτε. Τέλος. εσείς απαξιώνετε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τόσο στη χώρα σας όσο και εκτός. Και υπάρχει μια αρχή που εγώ ως πολιτικός έχω πάντα στο νου μου. Πρέπει να είναι κανείς καλός απέναντι στους ανθρώπους, γιατί κάποια στιγμή θα τους χρειαστεί. Ευχαριστούμε κυρία Γιουρόκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή ότι η έκθεση αυτή είναι γεμάτη ψέματα και παραπληροφόρηση και να ξέρετε ότι πολλά από αυτά που λέει η έκθεση αυτή έχουν να κάνουν με την προηγούμενη κυβέρνηση και όχι με την τωρινή του κ. Ορμπάν. Μιλάτε για παραστρατιωτικές ε, δυνάμεις που τρομοκρατούν τον κόσμο στα χωριά. Αυτά ήταν πριν το 2010, όταν ε, ήταν εκεί οι σοσιαλιστές. Και όντω τρει-τέσσερι μήνε έκαναν ε, τέτοια προεκλογική εκστρατεία οι σοσιαλιστέ, οπότε δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Σαρτζετίνη λέει ότι ήλεγξε ξανά και ξανά τα όσα αναφέρει στην έκθεσή της. Και πάλι όμως εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που αναφέρετε. Εγώ ποτέ δεν άκουσα για παραστρατιωτικές δυνάμεις, ναζιστικές στη Σουηδία κτλ. Εσείς κατηγορείτε ε, τι γίνεται με τους Ρωμά στην Ουγγαρία τώρα, αλλά όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση. Λέτε κάπου ότι, τα, ότι υπάρχει διάκριση σε βάρος των παιδιών των Ρωμά και ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί απέναντι στα παιδιά αυτά. Σύμφωνα όμω με έρευνε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν συγκρίνουμε την κατάσταση με το 2011, φαίνεται από την έκθεση αυτή ότι έχει μειωθεί ο αριθμό των παιδιών που αφήνουν το σχολείο, τον καταλείπουν. Ότι πάνε τα παιδιά αυτά στο σχολείο από την ηλικία των τρόνων γιατί έχει αλλάξει η νομοθεσία, λοιπόν έχει αλλάξει η κατάσταση. Τα παιδιά αυτά έξι χρονών μπορούν, έχουν μάθει αρκετά πράγματα για να μπορούν να μπουν στο κανονικό πια σχολείο για να το παρακολουθήσουν. Οπότε δεν μπορείτε να λέτε ότι η κατάσταση όσον αφορά τα παιδιά των Ρωμά έχει χειροτερεύσει. στα σημεία 46 και τα λοιπά λέτε επίσης ότι οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες που έχουν οι Ρώμα έχουν μειωθεί. Μα όχι, το αντίθετο συμβαίνει. Γιατί όλο και περισσότερα παιδιά Ρωμά πηγαίνουν συχνά στο σχολείο. Στο σημείο 45 επίσης λέτε κάτι ψέματα. Θα πρέπει να τα διορθώσετε αυτά τα σημεία. Αν τα διορθώσετε, αν μη τι άλλο, θα σώσετε κάπως την επαγγελματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί η σημερινή συζήτηση θα σοκάρει τους Ευρωπαίους πολίτες αν τα διαβάσουν αυτά. Και ζητάω από τη γραμματεία να μου πει πώς είναι δυνατόν αυτή η έκθεση να περιλαμβάνει τέτοιε παραγράφους, τέτοια σημεία, τα οποία τότε δεν είναι αλήθεια. Πώ γίνεται. Πώ γίνεται να γνωρείτε πλήρω τι δικέ μα παρατηρήσει κατά τη σύνταξη τη έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ για δύο λεπτά. Η επόμενη. Κυρία Κουτζίσικα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να απευθυνθώ στους Ούγκρους συναδελφούς και στον κύριο Υπουργό θα ήθελα να σας πω ε, να κοιμηθείτε καλά το βράδυ και να ξαναδιαβάσετε την έκθεση και μετά θα δείτε ότι η έκθεση της κυρίας Σαρτζεντίνη βασίζεται σε γεγονότα. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, να μην ε, θεωρείτε ότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα παιχνίδι και κάποιος ε, πρέπει να κερδίσει έναντι κάποιου άλλου εμείς ε, είχαμε συμφωνήσει στο να ε, μοιραστούμε τέτοιες αξίες ε, στο παρελθόν. Τότε είχαμε συμφωνήσει με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες. Στο παρελθόν ήμασταν υποκομμουνιστικό καθεστώς και τότε αυτές οι οργανώσεις ε, ήταν ε, πάρα πολύ επιτυχείς στην καταπολέμηση του κανονισμού και τώρα μάλιστα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν σας αρέσουν αυτές οι οργανώσεις. Λέτε ότι όλες αυτές οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις και ο όρος λένε ψέματα. Όμως θεωρώ ότι οι δράσει σας θα σημαίνουν ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το έθρο 7 συν το χρόνο ή θα παγώσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή θα περικοπούν σημαντικά για τη χώρα μας. Και επομένως ε, θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη στη χώρα. Έτσι λοιπόν θα μας ε, οδηγήσετε στο να είμαστε πολύ γρήγορα υπό την επιρροή του Πούτιν. Ξανασκεφτείτε λοιπόν, παρακαλώ αυτά που λέτε, ξαναδιαβάστε την έκθεση και μην θεωρήσετε ότι η συζήτηση αυτή καταφέρεται εναντίον σας ή κατά της ουγγρικής κοινωνίας. Θέλουμε η Ουγγαρία και όλη η Κεντρική Ευρώπη να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε στενοί εταίροι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 206 μπορούμε να δώσουμε το λόγο το πολύ σε δύο ε, μη μέλη της Επιτροπής, αλλά θα μιλήσουν μέχρι ένα λεπτό η κυρία Μορβάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή χάρη στις δικές σας επιθέσεις έχει αυξηθεί η εθνική συνοχή. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όλοι όσοι μας ακούν θεωρούν ότι είναι πολύ καλό να είναι Ούγγροι. Και επίσης ε, μας έχουν ε, ευχαριστήσει επειδή περασπίζουμε την εθνική κυριαρχία κατά της μετανάστευσης μας. Δίνετε την ευκαιρία ο κόσμος να δει τις προσπαθίες μας και να τις αναγνωρίσει. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Θέλω να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτίθεται εδώ στην Ουγγαρία και στην Πολωνία δύο χώρες που στην πραγματικότητα θέλουν με τη μεγαλύτερη υπεποίθηση να είναι στην Ευρώπη. Φυσικά όλα αυτά γίνονται επειδή προετοιμάζετε τις επόμενες ευρωεκλογέ ε, και ε, σίγουρα η σύνθεση αυτού του κοινοβουλίου δεν αντικατοπτρίζει καθόλου τις πεπιθήσεις των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Θα πρέπει να αλλάξει. Και αν ε, δεν υπάρχει πλέον ε, αυτό το λαϊκό κόμμα θα πρέπει να γίνει ένα καινούριο έτσι ώστε και στην επόμενη θητεία να ε, εκπροσωπούνται οι αξίες της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τσεβέρ. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα μέλη του ΕΛΚ δεν έχουν την ίδια άποψη. Είμαστε πολλοί που έχουμε διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό. Επομένως, ε, η συζήτηση αυτή δεν είναι πολύ καλή. Δεν νομίζω ότι ενδυναμόμουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση ε, Ορμπάν έχει κάνει πολλά για την ένταξη των Ρωμά αλλά και άλλων μειονοτήτων. Παραδείγματο χάρη, πριν λίγα χρόνια η σλοβενική μειονότητα ήταν στα όρια τη εξαφάνιση στην Ουγγαρία. Όμω τώρα με τη βοήθεια τη ουγγρική κυβέρνηση ε, είμαστε και πάλι ισχυρό εταίρο. Τα ξέρω αυτά τα θέματα γιατί είμαστε γειτονική χώρα με την Ουγγαρία. Έτσι λοιπόν δεν θα ήμουν τόσο κάθετος ε, σε όλες αυτές τις κατηγορίες που αναφέρονται στην έκθεση κατά της κυβέρνησης στην Ουγγαρία. Επίσης, ε, θέλω να πω ότι θα πρέπει να τους σεβόμαστε περισσότερο τους υπολείπους εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσει ο υπουργό, όπως είχαμε συμφωνήσει. Πέντε λεπτά το πολύ παρακαλώ. Και μετά την κυρία Σαντζεντίν. Μία ερώτηση μερικές ε, μήκοι όμικρον είναι σε κατάσταση ανάγκης και η κοινωνία των πολιτών ανησυχεί. Είπατε ότι υπάρχουν 65.000 ε, μήκοι όμικρον που, κυκλοφορούν στην, που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία σήμερα. Γιατί φοβάται η κυβέρνηση την κριτική από τις οργανώσεις αυτές γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την κριτική. Γιατί ασκείτε πιέσει αυτή τη ΜΚΟ, στη ΜΚΟ ε, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών. Γιατί τις πιέζετε να φύγουν ή να σταματήσουν να λειτουργούν. Αυτή είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με την έκθεση της κυρίας σας, γιατί αρνείστε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, η διεθνή Αμνηστία. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Καλά δεν αισθάνεστε αρκετά δυνατοί για να αντιπαρατεθείτε στην ε, Διεθνή Αμνηστία. Σε όλες τις άλλες χώρες της υπάρχει ισχυρή κοινωνία των πολιτών που πολλές φορές ε, έχει ε, διαφορές απόψε με την κυβέρνηση. Παρακαλώ πέντε λεπτά. Αξιότιμα μέλη. Με βάση αυτά που άκουσα, δεν μπορώ παρά να εξάγω το εξή συμπέρασμα το να επιτίθεστε κατά της Ουγγαρίας φαίνεται ότι είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό από σας. Το να ε, συκοφαντείτε την Ουγγαρία είναι κάτι το οποίο το θεωρείται φυσιολογικό και το να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας αυτό δεν το θεωρείται φυσιολογικό. Οποιοςδήποτε σέβεται τη δημοκρατία δεν θα μπορούσε να δεχθεί την προσέγγιση σας. Πρόεδρος. Κοιτάξτε. Κάποια μέλη χρησιμοποίησαν ε, αρκετά ε, έντονα φορτισμένο λεξιλόγιο και τρόπο Σα Παρακαλώ σε αυτό το πεντάλεπτό σα, Εντάξει, έχουν περάσει 30 δευτερόλεπτα. σα παρακαλώ ε, να θυμηθείτε ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια και σοβαρότητα. σα παρακαλώ να χρησιμοποιείτε τρόπο έκφραση που να αρμόζει στην αξιοπρέπεια του κοινοβουλίου. Τουλάχιστον προσπαθήστε. Κοιτάξτε. Εξετάζουμε την έκθεση κυρία Αργεντίνη. Αυτό είναι το θέμα. Αν μπορείτε να σχολιάσετε τον τρόπο παρουσίαση τη έκθεση. Δεν θα ήθελα να υπάρξει μεγάλο ακόμα. Παρακαλώ, συγκεντρωθείτε στα συγκεκριμένα θέματα που θέτει η κυρία Αργεντίνη και τις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, νόμιζα ότι υπήρχε ελευθερία έκφραση εδώ μέσα. Ελευθερία έκφραση γνώμη και ότι ισχύει και για μένα σε αυτό το σώμα. Αν δεν ισχύει, θα συμμορφωθώ με τις αποφάσεις σα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εδώ, κατά τη συζήτηση, ε, έχει κατασκοφαντηθεί η Ουγγαρία. Και δεν μπορώ να δεχθώ να μου υπαγορεύετε πώς θα απαντήσω. Και εγώ, όπως και εσείς, δίνω τη γνώμη μου για αυτά που υπόθηκαν. Κοιτάξτε, υπενθυμίζω. Έχουμε κερδίσει τρεις συναπτές εκλογές με πολύ ευρείες πλειοψηφίες γιατί με ρωτάτε ε, σε τι βαθμό νομιμοποιούμε να εκπροσωπώ τους Ούγγρους. Θα μπορούσα και εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Σας ρωτήσω πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες ε, σας εξουσιοδότησαν ε, να κάνετε μαθήματα εδώ στο λαό της Ουγγαρίας. Και απευθύνονται και κατηγορίες για τον αντισημιτισμό. Στην Ουγγαρία συζητάμε με τον Γιώργη Σόρος. Μπορεί να μην συμφωνούμε, ιδιαίτερα για τα θέματα μετανάστευσης. Αλλά, ε, όπως ξέρετε, ο, ο κύριος Σόρος, ε, και δεν το έκρυψε, δεν ήθελε να κερδίσουμε εμείς τις εκλογές. Όταν συζητάμε με τον κύριο Σόρος, δεν εξετάζουμε τη θρησκεία του ή τις απόψεις του γενικότερα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ένας πράσινος ευρωβουλευτής, ο οποίος έφυγε εκ τότε, μας κατηγόρησε και το Ιόμπικ, το ακροδεξιό κόμμα, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προεκλογική τους εκστρατεία, οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές δηλαδή, είχαν ένα μόνο θέμα στην προεκλογική τους εκστρατεία. Πώς θα μπορέσουν να συνάψουν συνασπισμό με το ΙΟΜΠΙΚ για να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Και τώρα εσεί κατηγορείτε εμένα ότι συνεργάζομαι με αυτό το ακροδεξιό κόμμα. Οι σοσιαλιστέ και οι πράσινοι αυτό έκαναν κατά την προηγουμένη εκστρατεία ακριβώ. Επίση, να έχετε υπόψη σα. Έχουμε αποστείλει τεκμηριωμένες απορρίψεις όλων των θεμάτων που θέτει η έκθεση και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα σας απαντήσω ως εξής. Ο Ουγγρικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να προϋποθέτει και να απαιτεί διάφανη χρηματοδότηση των οργανώσεων που επιδιώκουν να επηρεάσουν την Ουγγρική κοινή γνώμη. Είναι λογικό να αναμένεται διαφάνεια, για παράδειγμα, από τα πολιτικά κόμματα. Άρα εξίσου λογικό να υπάρχει και η ανάλογη διαφάνεια από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και που θέλουν να παίξουν ένα ρόλο στην ουγγρική πολιτική σκηνή. Γιατί να κρύβουν ποιος τους χρηματοδοτεί. Και κύριε Πρόεδρε. Εξανίσταμε και για αυτό που είπατε ότι δεν επιτρέπουμε στις ε, ΜΚΟ να λειτουργήσουν στην Ουγγαρία. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι οι ΜΚΟ όμικρον να γνωστοποιούν τους χρηματοδότες τους. Αυτό δεν δυσχεραίνει την λειτουργία τους. Γιατί να μην βάλουν στο site τους ποιοι τους χρηματοδοτούν. Αυτή είναι η γνώμη μας και θα εμείνουμε ότι η διαφάνεια είναι σημαντική. Τώρα, η ελευθερία της πανεπιστημιακής κοινότητας. Έχουμε πάνω από 20 ξένα πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Ουγγαρία. Το μόνο που διαμαρτύρεται για το νέο νόμο είναι το Πανεπιστήμιο της ε, Κεντρικής Ευρώπης. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία Αμερικανικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Ουγγαρία. Και ακούτε μόνο τα παράπονα ενός και μόνου. Γιατί αφού μπορούν να λειτουργήσουν και είναι δεδεθειμένα να λειτουργήσουν και είναι δεδεθειμένα να υπογράψουν σύμφωνα συνεργασία με ένα το Μέριλαντ αυτό το πανεπιστήμιο, γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Χαίρομαι ιδιαίτερα και εκτιμώ το ότι μου δώσατε δυνατότητα να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας, αλλά εξακολουθούμε να καταδικάζουμε το ότι διαδίδεται ψέματα κατά της Ουγγαρίας. και θα σας στείλω και τεκμηριωμένη γραπτή απόρριψη όλων των σημείων που φέρετε στην έκθεση, αλλά ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Ευχαριστώ και τον λέει ο Πρόεδρο που μα επιτρέπουν να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Και τώρα η συγγήτρια, η κυρία Σαρτζεντίνη, για να ολοκληρώσει και να κλείσει. Διαδικαστικό έχετε. Αν είναι διαδικαστικό παρόλο να είναι. Μόνο διαδικαστικό, έτσι. Αν είναι διαδικαστικό θα σας διακόψω. Είναι διαδικαστικό, αλλιώς θα σας διακόψω. Hm. Αν δεν είναι διαδικαστικό θα σας διακόψω. Η Γενική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ο σεβασμός των μειονοτήτων. Οπότε, Πρόεδρε, σας ζητώ να προστατεύσετε την άποψη των μειονοτήτων στην αίθουσα αυτή. Γιατί εδώ πρόκειται για μία επίθεση. Έχουμε το δικαίωμα να εκφραστούμε ως μειονότητα. Και σας ζητώ να προστατεύσετε την ελευθερία της εργασίας μας εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Κύριε Σαρτζεντίνη, συνεχίστε παρακαλώ. Μας δώσανε χρόνο οι διερμηνείς, οπότε μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς, λέει η συγγήτρια. Κύριε Σαρτζεντίνη, σε μια συζήτηση σαν κι αυτή, όπου φαίνεται σαν να μην μιλάμε μεταξύ μας, καλό θα ήταν να μπορεί κανείς να τοποθετηθεί με σωστή γλώσσα. Λοιπόν, σε αυτούς που λένε ότι υπάρχουν σφάλματα στην έκθεσή μου, παρακαλώ να τα διορθώσετε. Αν νομίζετε ότι έχω κάνει λάθη, με τροπολογίες μπορείτε. 15 του μηνός, 15 Μαΐου, αν δεν απατώμενη η προθεσμία. Πρόεδρε, οι ευρωβουλευτές βέβαια κάνουν πολιτική και εγώ. Εδώ όμως μου ανατέθηκε η κατάρτιση μιας έκθεσης από την Ολομέλεια και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να είμαι ανοιχτή σε διάφορες απόψεις και να μην μεροληπτήσω καθόλου. Οπότε αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι παρόλο που είμαι τόσο ευγενή, που επιτρέπω στην Ουγγρική κυβέρνηση να έρθει ξανά και ξανά να εκφραστεί, αναμένω, αν μη τι άλλο από την ε, Ουγγρική κυβέρνηση, να συμπεριφερθεί κυβερνητικά. Δεν μιλάω σε ένα πολιτικό κόμμα. Μιλάω σε έναν υπουργό που εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Το να μπερδεύουμε το κόμμα, την κυβέρνηση, το κράτος και το λαό, αυτό είναι κάτι το οποίο επανέρχεται ξανά και ξανά στις συζητήσεις μας. Φυσικά και είσαστε ελεύθερος να έρθετε να μιλήσετε και να πείτε ό,τι θέλετε και ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να πείτε. Όμως μπορώ να παρατηρήσω ότι με εκπλήσει που στην Ουγγαρία ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στρεβλώνει τα όσα λέω και χρησιμοποιεί το όνομά μου λέγοντας ότι ψεύδομαι. Στη δικιά σας έκθεση που μας στείλετε, όπου προσπαθείτε να αντιδράσετε στη δικιά μου έκθεση, λέτε ότι η συγγήτρια σαφώς δεν βασίζεται στις δικές της έρευνες, στους διάφορους τομείς πολιτικής και τα συμπεράσματά της δεν είναι δικά της. Ναι, πράγματι μελέτησα. Μελέτησα την πληροφορία και αυτή την πληροφορία που μελέτησα και την πήρα από διάφορους οργανούς τη χρησιμοποίησα. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι ψεύδομαι. Και μετά να λέτε ότι καμία από τις πληροφορίες που χρησιμοποίησα ε, δεν ε, απορρέει δικά μου συμπεράσματα δεν είναι σωστό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει η συζήτηση που κάνουμε εδώ να σέβεται τους πάντες. Το επόμενο στάδιο είναι η διαδικασία υποβολής τροπολογιών. Όπως είπα και στην αρχή, εδώ δεν κάνουμε διαπραγματεύσεις με μια χώρα μέλος, πρόκειται για μια έκθεση η οποία πρέπει να καταλήξει στα χέρια του Συμβουλίου. Και αυτό κάνω με όλους τους συναδέρφους που είναι σκιώδεις εισηγητέ. Οπότε προσβλέπω στις δικές σας προτάσεις τροποποίησης εφόσον υπάρχουν. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 15η Μαου, συνάδελφοι, στι 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ όλου του συναδέρφους για τη συμμετοχή σα στη συζήτηση εδώ.